Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του 2018 για την Επιτροπή μας. Την Επιτροπή μας, την Υποεπιτροπή Άμενας και Ασφάλειας. Τα περισσότερα μέλη από την Πολωνία βρίσκονται εδώ, γι' αυτό το λόγο επιλέγω τη μητρική μου γλώσσα για να ξεκινήσω τη συνεδρίες και θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά σε όλου. στην αρχή αυτή της διήμερη συνεδρίασης. Θέλω να σα υπενθυμίσω σε όλους ότι όπως συνήθως η συνεδρίασή μας αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τη διερμηνία, η προτεραιότητα στη διερμηνία δίδεται στις γλώσσες των ε, μονίμων, των τακτικών μελών της Επιτροπής. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης, ε, στην ε, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν σχόλια... Θα θεωρήσουμε ότι η ατζέντα, ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Έχουμε και την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 22ης και 23ης Νοεμβρίου του 2017 καθώς και των πρακτικών της 7ης Δεκεμβρίου του 2017. Αν έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές, έχετε χρόνο μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ε, αυτής της ε, Υποεπιτροπής ε, Ασφαλείας και Άμενας, δηλαδή μέχρι την ώρα του μεσημεριανού αύριο. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Θα πρέπει σήμερα να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 5 και 4. Λίγο νωρίτερα από τη συνήθως. Κάποια σημεία στην ημερήσια διάταξη ε, είχαμε, εκ των οποίων ένα αφορούσε μια ανταλλαγή απόψεων για το Brexit με τον ε, εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις ε, ε, ενός άλλου εμπειρογνώμουνα. Ωστόσο, ένας από τους συντονιστές είπε πάρα πολύ σωστά και μετά από διαβούλευση με τη γραμματεία αποφασίσαμε να αναβάλουμε το σημείο αυτό. διότι και εγώ και ένας δυο συντονιστές ε, θα πρέπει να παραστούμε σε μια ε, συμβουλευτική συνεδρίαση με την ε, Διαχειριστική Επιτροπή όπου θα συζητήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με το Brexit, την ασφάλεια και την άμενα. Οπότε θα κλείσουμε στις 5 και 4. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σημερινή ημερησία διάταξη και με μεγάλη μου χαρά και τιμή για άλλη μια φορά φιλοξενώ τον πρόεδρο της Στρατιωτική Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον στρατηγό Μιχαήλ Κωνσταράκο, που είναι γνωστό σε όλους σας, σε όλους μας. Είναι ο πρόεδρος ε, του ανώτατου ε, στρατιωτικού οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η χρονιά ε, είχε χαρακτηριστική από πολλές εξελίξεις στον τομέα της κοινή πολιτικής ε, ασφαλείας και άμυνας ε, με πολλά πράγματα που συζητήθηκαν εκτενώς στο Συμβούλιο και τόσο και από τις Επιτροπές ΕΝΤΕ, ΑΦΕΤ, στην Ολομέλεια, στις διάφορες συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδήγησαν όλα αυτά στην έγκριση πολλών σημαντικών εκθέσεων. Όλοι μας λοιπόν ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε τις απόψεις του στρατηγού Μιχαήλ Κωνσταράκου για τις ε, επιχειρησιακές ε, αλλαγές ε, που έχουν γίνει και για τις προοπτικές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των κρατών μελών σε αυτό το τομέα. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις και είμαι βέβαιη ότι και οι συναδελφοί μου θα έχουν ερωτήσεις όσον αφορά τις ε, δικές σας δραστηριότητες ε, στρατηγέ. Παρατήρησα ότι τελευταία επισκεφθήκατε ε, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 χώρες όπως το Βιετνάμ. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να μάθουμε ποιες είναι οι εξελίξεις στην από Ανατολή. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις ε, όσον αφορά τις προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και που αντιμετωπίζουμε ήδη εδώ και κάποιο καιρό. Χωρίς άλλη καθυστέρηση δίνω το λόγο στον στρατηγό κύριο Κωνσταράκο. Έχετε το λόγο. Madam Chair. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πριν ε, προχωρήσω με την ομιλία μου, θέλω να ευχηθώ σε εσά και στου συγγενεί σα ε, τι καλύτερε ευχέ μου για ένα ευτυχέ και επιτυχέ νέο έτο και ελπίζω όλε τι προσπάθειε ε, να ευοδοθούν. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μεταξύ των ερετών εκπροσώπων ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεγάλη μου χαρά έχω την ευκαιρία να σα ενημερώσω για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής ε, στην ε, κοινή ε, πολιτική ασφαλείας και άμενας. Κυρίες και κύριοι, πριν από δύο χρόνια, όταν ήρθα στην Επιτροπή αυτή, ολοκλήρωσα στο τέλος λέγοντας ότι καθώς μιλάμε σε πολλές περιοχές του κόσμου η αστάθεια εντείνεται και ότι πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή και ενωμένοι παρά τις διαφορές μας. Μέσα σε αυτή τη διετία που έχει παρέλθει, ο κόσμος δεν έγινε πιο ασφαλής, ούτε πιο σταθερός οποιαδήποτε πρόοδος στον τομέα της ασφάλειας, ε, το κοινό σχέδιο δράσης, ε, η ε, συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν συνοδεύτηκαν και από την υποβάθμιση των σχέσεων αλλού, όπως στην Βόρειο Κορέα και στην Ιεμένη. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις και οι δράσεις της οι κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα αλλάζουν. Αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπου. Ε, ε, με το απεσιόδοξο σενάριο ότι αποτύχαμε στου στόχου μα και ότι συνεπώ ε, παραμένουμε στι χώρε αυτέ. Ο άλλο τρόπο ερμηνεία είναι ο αισιόδοξο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται αξιόπιστο πάροχο ασφαλεία και του ζητείται συνεπώ να παρέχει υποστήριξη παρά του περιορισμού που υπάρχουν. Και οι δύο πτυχέ φυσικά είναι σωστέ. Θα επιστρέψω στο ζήτημα των επιχειρήσεών μας και των δράσεών μας αργότερα στην παρουσίασή μου. Στην ε, απόφαση του Συμβουλίου της 22ης ε, Ιανουαρίου του 2001 με την οποία συστήθηκε η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρει την αποστολή τη ως εξή. Η Στρατιωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για να παρέχει στην ε, Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας ε, συμβουλές στρατιωτικές ε, για όλα τα στρατιωτικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει τις στρατιωτικές κατευθύνσεις για όλες τις δραστηριότητες εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με αυτή την αποστολή η Στρατιωτική Επιτροπή δραστηριοποιείται ενεργά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα σε όλα τα επίπεδα συμμετείχε στην εκπόνηση της ε, συνολικής ε, στρατηγικής στρατηγικής από την αρχή. Ε, λήφθηκαν υπόψη τα σχόλιά μας και υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίστηκε οι θέσεις μας ότι η ασφάλεια και η άμυνα έχουν γίνει βασικά ζητήματα για τους ευρωπαϊκούς λαούς και ότι αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και να αντιμετωπίσετε στο γενικότερο αυτό Ευρωπαϊκό Έγγραφο Στρατηγική. Γνωρίζουμε τώρα ότι η άμυνα και η ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο τη παγκόσμια στρατηγική και ότι επηρεάζουν όλα τα ε, έγγραφα που προκύπτουν. Με αυτή μας τη συμμετοχή στην ε, φάση σχεδιασμού και υλοποίησης και βάσει της συμβολής μας ε, στην Παγκόσμια Στρατηγική, εμείς ως Στρατηγική Επιτροπή εξακολουθούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες συστάσεις και συμβουλές στους συντάκτες του σχεδίου υλοποίησης βάσει της τεράστιας στρατιωτικής εμπειρίας που έχει ο οργανισμός μας. Θα γνωρίζετε φυσικά ότι η φάση υλοποίηση ήταν το αμέσως επόμενο βήμα, χωρίς ενδιάμεσο βήμα, ούτε λευκές βίβλους, ούτε τίποτα άλλο. Η Επιτροπή επίσης συμμετείχε σε διαφορετικό επίπεδο στην εκπόνηση των παραδοτέων του σχεδίου υλοποίηση. δηλαδή την δομή, τη μόνιμη δομή συνεργασία στην ΠΕΣΚΟ, τη συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση της άμυνας που είναι γνωστή ως κάρτα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Αυτή η συμμετοχή στην φάση σχεδιασμού δεν ε, ολοκληρώνει τη συμβολή μας. Αντιθέτως, η Επιτροπή μας ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συμμετοχή μας και στη φάση υλοποίηση. Στις θέσεις των κρατών μελών που εκφράζονται μέσω της, Επιτροπής, της Στρατηγικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρεται ότι απαιτείται εκτενή συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η πολιτική διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές γνώσεις που μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικές συμβουλές στρατιωτικές που θα ενταχθούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό λαμβάνεται υπόψη και αποτυπώνεται στα έγγραφα που καθερώνουν τις ε, διαδικασίες μέσω των οποίων ε, θα εργάζονται όλες, όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Σε όλα τα έγγραφα που έχουν εκπονηθεί μέχρι στιγμής ε, τελικά και σχέδια προβλέπετε κάποιους ρόλους για τη Στρατιωτική Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία τη συμβολή τη. Για τα έργα ΠΕΣΚΟ, ο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2017, τον Νοέμβριο αναφέρεται ότι η Στρατιωτική Επιτροπή θα παρέχει ε, στρατιωτικές συμβουλές για στρατιωτικά προγράμματα και εμείς παρέχουμε στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας στρατιωτικές συμβουλές και συστάσεις όσον αφορά ε, την ετήσια ε, διαδικασία αναθεώρησης της ΠΕΣΚΟ. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα παίξει η Στρατιωτική Επιτροπή στις διαδικασίες οι οποίες θα καθιερωθούν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας. Όπως καταλαβαίνετε εδώ η θέση της ε, Στρατιωτικής ε, Επιτροπής θα ενταχθεί. Η συμμετοχή της μαζί με όλους τους ενδιαφερομένους ώστε να εντοπιστούν οι βέλτιστοι τρόποι χρονικά και απόψη και μεθοδολογικά ώστε να συντονιστούν οι απόψεις τους ε, και να συμμετέχει σε όλες τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτή τη φάση πρέπει να υπογραμμιστεί κυρίε και κύριοι ότι η Στρατιωτική Επιτροπή ανέκαθεν συμμετείχε σε στρατηγικό επίπεδο στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ακόμη και πριν από τα τελευταία γεγονότα. Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά ε, στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων για την διατήρηση, τη βελτίωση ε, και την κάλυψη των νέων αναγκών στο πλαίσιο της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Έτσι εκπονήθηκε ο κατάλογος απαιτήσεων, παρέχονται ε, οι διάφορες απαιτήσει στρατιωτικών ικανοτήτων που τροφοδοτούν ε, τα σχετικά σχέδια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2016, οι νέε φιλοδοξίε που παρέχει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν τη Στρατιωτική Επιτροπή να υιοθετήσει το νέο κατάλογο απαιτήσεων βάσει των διαφόρων σενάριων. Αυτό οδήγησε στην αναθεώρηση των ε, του καταλόγου απαιτήσεων που είχε συνευθεί τον Νοέμβριο του 2017. Αποτελεί του τους θεμέλιους λίθους ε, μαζί με τους άλλους ε, καταλόγους για το σχέδιο στρατητικής ανάπτυξης. Οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων καταλόγων και σχεδίων είναι προφανείς, δεν χρειάζεται να τους αναλύσω. όλα τα διαφορετικά επίπεδα και οι διάφοροι τρόποι συμμετοχή ε, στην κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα ε, μα ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον. Η συμμετοχή όμω τη Επιτροπή εστιάζεται και στο παρόν. Με έξι τρόπου βελτίωση τη απόδοση των επιδόσεων ε, του στρατιωτικού σκέλου. Ε, θεωρείται σημαντικό στοιχείο ε, για την συνολική προσέγγιση ε, της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξωτερικές συγκρούσεις. Την ονομάζουμε σήμερα ολοκληρωμένη προσέγγιση επίσης. Θέλουμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή της. Για το σκοπό αυτό θεωρώ την καθιέρωση ε, της μονάδας σχεδιασμού και στρατιωτικών ικανοτήτων ε, σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για τη βελτίωση ε, της ε, των στρατικών δυνατοτήτων. Εμείς επιμένουμε να τονίζουμε τα κενά που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής ηγεσία επιτόπου στις επιχειρήσεις συστάσεις που έχουν γίνει, έχουν υιοθετηθεί και υλοποιηθεί. Επίσης δημιουργήθηκε και ένα αρχηγείο για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το οποίο από στρατιωτική άποψη δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Ελπίζουμε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις συστάσεις ε, της αναθεώρησης που προβλέπεται να λάβει χώρα πριν από το τέλη του έτους. Σε τακτικό επίπεδο η Στρατιωτική Επιτροπή ε, διευθύνει όλε τι στρατιωτικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στη φάση σχεδιασμού και εκτέλεση ε, των στρατιωτικών επιχειρήσεων και δράσεων στο πλαίσιο τη κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα. Θα σα παρουσιάσω εν συντομία την ε, κατάσταση των έξι σημερινών επιχειρήσεων και δράσεων. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή Εκπαίδευση στη Σομαλία ξεκίνησε το 2010 βάσει μια προσέγγιση τριών σκελών. Εκπαίδευση, συμβουλέ και καθοδήγηση βοηθά τις αρχές της Ομαλίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση ειδική ε, εκπαίδευση μέσω μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ε, στρατόπεδο Αλτζαζίρα στο Ιλμογκαντήσου. Μέχρι στιγμής ε, η επιχείρηση αυτή έχει εκπαιδεύσει περίπου 5.500 Ομαλούς στρατιώτες. Η συμβουλευτική ομάδα της αποστολής παρέχει στρατηγικές συμβουλές στις ε, Σομαλικές Αρχές μαζί και στο Υπουργείο Άμυνα και στο Γενικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλέ προκλήσει. κύρια είναι η πρόσφατη προσπάθεια της Ομαλικής Κυβέρνησης να ενισχύσει την αρχιτεκτονική της εθνικής ασφάλειας και οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις από το στρατό της Ομαλίας με την υποστήριξη άλλων ενδιαφερομένων επίσης όπως της ε, ε, αποστολής Αφρικανικής Ένωσης στην Σομαλία. για την καταπολέμηση των διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων που ε, λιμένονται στη χώρα. Αυτές οι προκλήσεις δίνουν τη δυνατότητα στην αποστολή μας να ενισχύσουμε την υποστήριξη ε, στην, όσον αφορά την εκπαίδευση του Σομπαλικού στρατού και την παροχή συμβουλών σε στρατιωτικά θέματα. Επίση, υπάρχουν και διάφορε ανησυχίε όσον αφορά την κατάσταση ασφαλεία στη Μογκαντήσου και την απειλή τη Αλσαμπάμπα. Θα βλέπετε πολλά από αυτά ε, τα περιστατικά σίγουρα στι ειδήσει. Αυτά όσον αφορά την πολιτική ε, αστάθεια στη Σομαλία. Μετά έχουμε την ε, εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλί που ξεκίνησε το 2013 και στέθηκε με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές δυνάμεις του Μάλι ε, αντιμετωπίζουν υπερβολικά πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν και η αποστολή μας εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα. Η συνολική αξιολόγηση του συμβουλευτικού σκέλους επίσης είναι θετική. Επίσης ε, ανέλαβε ένα νέο στόχο να συμμετέχει η αποστολή μας ε, ε, στις δυνάμεις του G5 Sahel ενισχύοντας τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο των εθνικών δυνάμεων G5 Sahel. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο Μάλι είναι η περιφερειακή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιφέρεια σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων του Μάλι, η ευελιξία που απαιτείται για... ώστε οι στρατιωτικές δυνάμεις ε, να αντιμετωπίσουν το μέλλον, να προετοιμάσουμε δηλαδή μέσω εκπαίδευση τις στρατιωτικέ δυνάμεις και η βαθμία πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας στο Μάλι. Αυτά που μα ανησυχούν είναι η αναδυόμενη ριζοσπαστικοποίηση και ε, στρατολόγηση στη βόρεια περιοχή της χώρας ε, η κατάσταση στον Παμάκο και στον ΚΑΟ, η πολιτική αβεβαιότητα ε, καθώς κινούμαστε προς εκλογές ε, και η εφοδιαστική αλυσίδα και η σχετική υποστήριξη. Η κεντροαφρικανική δημοκρατία, η αποστολή μας έχει μετατραπεί σε εκπαιδευτική. Και εδώ η αποστολή μας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. πιο σημαντική είναι η εκπαίδευση επιπλέον προσωπικού στο πλαίσιο ε, της διαδικασίας DDR, αποστρατικοποίησης ε, και μεταρρύθμισης. Η υπόθεση των μονάδων ΦΑΚΕ στην χώρα που είναι ο Εθνικό Στρατό, οι ανησυχίε μα ε, αφορούν την πολιτική αστάθεια και την απειλή των στρατιωτικών ομάδων που δεν εμπλέκονται στη διαδικασία DDR. Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν ε, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μέσω τη συνεργασία των διαφόρων ενδιαφερομένων εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε εκεί μια ιστορία επιτυχία. Πάμε τώρα στι αποστολέ. Ε, από τι αποστολέ ε, στι εκτελεστικέ επιχειρήσει, η επιχείρηση Ανθέα στη Βοσνία Ερσεγοβίνη παρέχει εκπαίδευση διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τη χώρα από το 2004. Η κύρια προσπάθεια της ε, αποστολής αυτής είναι η εκπαίδευση των στρατιωτικών δυναμών της χώρας. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Έχουν αναπτυχθεί καλύτερες επαφές μεταξύ της αποστολής και του Γενικού Επιταλείου του Σεράγεβο ε, επειδή συνεργαζόμαστε ε, στην εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων. Οι υπερβολικά εθνικιστικέ οργανώσει, οι ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις και οι λοιπές απειλητικέ οργανώσει παραμένουν απειλή για την σταθερότητα τη χώρα και για την εσωτερική ασφάλεια. Απαιτείται μεγαλύτερη ε, επαγρύπνηση. Όσον αφορά τις υπόλοιπες προκλήσεις, ε, σημειώνονται οι εξή. Η ικανότητα της επιχείρησης Ανθία να ανταποκριθεί στις απειλές στο περιβάλλον αυτό ε, αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα. Η έλλειψη πληροφοριών και οι περιορισμένες δυνάμεις που υπάρχουν επί τόπου δεδομένου ότι είναι περιορισμένες οι εφεδρικές δυνάμεις που υπάρχουν εκεί. Αυτά που ανησυχούν εμένα, πέραν της πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα, σε σχέση με τις γενικές εκλογές που θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο του 2018 και την πρόοδο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επιβραδυνθεί το 2017 η Ευρώπη ιστορικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θάλασσα. Το ίδιο ισχύει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θαλάσσιος τομέας περιλαμβάνει ε, τη γραμμή ζωής της οικονομίας μας ε, και αυτό, έτσι δεν μας εκπλήσει ότι δύο από τις τρεις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θαλάσσιες. Στη Νότια και Κεντρική Μεσόγειο έχουμε ξεκινήσει την ε, επιχείρηση Γιούνα Φορμέτ Σοφία από το καλοκαίρι του 2015 ώστε να γίνουν συστηματικές προσπάθειες ε, συμβολή ε, στην διακοπή ε, της εμπορίας ανθρώπων και να πάψει η απώλεια ζώων στην Μεσόγειο. Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μεταναστών είναι μόνο μία πτυχή της προσπάθειας. Το να θέσουμε τέλος στην ανθρώπινη τραγωδία που παρατηρούμε να εκτελείστε στη Μεσόγειο θα αποτελέσει και σημαντική συμβολή για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή εντολή, η εντολή της επιχείρησης τροποποιήθηκε το 2017 και περιλαμβάνει πλέον και τις εξής, ε, ε, και εξής καθήκοντα. Ένα μόνιμο ε, μηχανισμό εκπαίδευσης ώστε να εκπαιδευτούν οι ακτοφυλακές νέες δραστηριότητες παρακολούθησης και συγκέντρωση πληροφοριών γιατί όλες τις παράνομες δραστηριότητες από τη Λιβύη σε συνεργασία με την UNHCR 246 και 262 και να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες ε, ε, κοινής χρήσης πληροφοριών ε, από όποια πηγή μπορούμε και τη Frontex και την Europol. Ε, κυρίες προκλήσεις θεωρώ ότι είναι η εξή. Η ενισχυμένη παρακολούθηση από τη Λιβική ακτοφυλακή και πιθανή εντολή δραστηριοποίησης εντός χωρικών υδάτων. Τέλος, Έχουμε τη Γιουναφόρα Ταλάντα, την πρώτη στρατιωτική θαλάσσια ε, ε, ε, επιχείρηση που ξεκίνησε το 2008 κατάφερε να εξαλείψει της, την πειρατική απειλή και βοήθησε στην ασφαλή παροχή πολλών τόνων φαγητού στα Σομαλικά λιμάνια. Τελείωσε τον περασμένο Μάρτιο και έκτοτε ξανά εμφανίστηκε η πειρατεία στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που υποστήριξα εγώ πριν από δύο χρόνια ενώπιον της Επιτροπής σας, ότι έχουμε εξαλείψει πολλές από τις δυνατότητες ε, της πειρατικής απειλής, αλλά όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα αποσύρεται, οι θαλάσσιες μονάδες που παρέχουν ασφάλεια στην περιοχή αποσυρθούν τότε ε, ε, εμφανίζεται ξανά η πειρατεία. Δεν είναι όλα όμως μαύρα. Η Unifor Atalanta έχει ε, δημιουργήσει σημαντικές σχέσεις συνεργασίας με διάφορους φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, τις διεθνείς θαλάσσιες δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, την Κίνα, την Κορέα, όλοι εμπλέκονται στην καταπολέμηση της πειρατείας. Η σπουδαιότητα της συνεργασίας που έχει γίνει με την ναυτιλία ε, παίζει σημαντικό ρόλο και επίσης ε, συνεργάστηκε η επιχείρησή μας με τη Σομαλία για να αναπτυχθούν θαλάσσιες δυνατότητες, ναυτικές δυνατότητες και με άλλα, άλλους φορείς. Ε, προκλήσεις θεωρώ ότι είναι οι εξής κυρίως το πώς επηρεάζει, επηρεάζουν οι συγκρούσεις ε, στην Ιεμένη, τις δραστηριότητες αυτές ε, και το πρόβλημα των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σομαλία και ειδικότερα για τις περιπτώσεις ε, διάσωσης και, και ένωσης σε περίπτωση εκτακτής ανάγκης. Όσον αφορά τις ανησυχίες για την κατάσταση αυτή, η πολιτική κατάσταση βρίσκεται σε πολύ υψηλή προτεραιότητα, όπως και ο εκτοπισμό των πληθυσμών. Όλα αυτά δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή μας στην εξέλιξη της κοινή πολιτική άμυνα και ε, ασφάλειας. Κοιτώντα προ το μέλλον, η ευθύνη μου να σας παρουσιάσω ιδέες και να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση για να την πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Στα δύο χρόνια της Προεδρίας μου έχουμε παράγει στο γραφείο μου πολλά έγγραφα και επιστολές με νέες ιδέες, με νέες πρωτοβουλίες που θεωρούμε ότι αξίζει να εξεταστούν ή να ειδωθούν με νέο μάτι. Πράγματα που έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, επειδή τώρα πλέον οι προϋποθέσεις, οι, οι συνθήκες έχουν οριμάσει και έχει έρθει η ώρα να τα ξαναδούμε με άλλο μάτι. Το ζήτημα που, τα ζητήματα που παρουσιάζονται σε αυτά τα έγγραφα είναι πολλά και διάφορα σε όλους τους τομείς, από την εξέλιξη των μάχημων ομάδων, μέχρι την ε, ισορροπία των φύλων, μέχρι την στρατηγική εκπαίδευση και την οικονομική αποζημίωση για ορισμένε περιπτώσει, καθώ και για τον ορισμό στρατητικών συμβολών στι ευρωπαϊκέ αντιπροσωπείε. Έτσι λοιπόν, ε, σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική Επιτροπή έχει δείξει δυναμισμό και πρωτοβουλία. Ε, τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με την πρωτοβουλία. Ορισμένες πρωτοβουλίες ε, αντιμετωπίζονται με ενθουσιασμό, άλλες ε, έχουν, ίσως είναι υπερβολικά πρωτοποριακές. Ε, εμείς προτείνουμε κάθε πρόταση και κάθε ιδέα να συζητείται με θετικό πνεύμα, χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Οι συζήτηση μας πρέπει να είναι πάντα ειλικρινείς, επικοδομητικές. Μια από τις πρωτοβουλίες που έγινε δεκτή με πολύ καλό μάτι ήταν η εκπαίδευση, ε, η σταδιακή εκπαίδευση για τη, σταδιακή, για τη σταδιακή δημιουργία της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Ταυτότητας. Το Ευρωπαϊκό Κολέγιο το Στρατιωτικό Κολέγιο έχει ε, προετοιμάσει το πρόγραμμα για το πρώτο έτος. Από την άλλη πλευρά, μια από αυτές τις πρωτοβουλίες που δυστυχώς ε, δεν πήγε καλά σχετιζόταν με τη χρηματοδότηση των μάχημων ομάδων. Οι μαχήμες ομάδες ε, ποτέ δεν ε, εστάλσαν σε επιχείρηση και αυτό μάλλον θα παραμείνει έτσι με στο ορατό μέλλον. Ο λόγος για τον οποίο απέτυχε αυτό το ε, εργαλείο που παρέχει πολλές δυνατότητες ήταν διτός. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε πολιτική βούληση και μετά υπήρχε υποχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Αθήνα. Η πρόσφατη αναθεώρηση του Μηχανισμού Αθήνα δεν ε, κάλυψε τις προσδοκίες μας. Εμείς θέλαμε απτή υποστήριξη για το μόνο εργαλείο ταχείας απόκρισης που έχει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία δεν ε, κατέληξε σε πραγματικές αλλαγές, αλλά μόνο σε ε, τμηματικές επιφανειακές θα έλεγα βελτιώσεις κάτι που δείχνει ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτό το τομέα στην ε, σκλήρη της εξουσία. Πρέπει να πω ειλικρινά ότι η σκληρή εξουσία, η στρατηγική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει ε, όχι επαρκώς αναπτυγμένη. Σε ένα τόσο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τόσο γρήγορο, η ύπαρξη ψευδών ειδήσεων ε, και οι επιπτώσεις των μηνυμάτων τρόμου και τρομοκρατίας προς πολίτες απαιτεί να είναι η Ευρώπη πάρα πολύ δραστήρια σε θέματα επικοινωνιών. Ε, οι προσπάθειε πρέπει να γίνουν από όλε τι πλευρέ. Εγώ, ω πρόεδρο τη ε, Στρατιωτική Επιτροπή, ω ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με άλλου αξιωματούχου, φοιτητέ, ακαδημαϊκού, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα στρατηγικά μηνύματα. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας αξιόπιστος, ισχυρός, ικανός και ειλικρινής και προβλέψιμος ε, πάροχος ασφαλείας. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους πολίτες και την επικράτειά της και ότι αυτή η ενίσχυση δεν πρέπει να θεωρείται απειλή κάτω οποιοδήποτε ε, πολίτη ή κράτους ότι η Στρατιωτική Επιτροπή θα παραμένει στο πλευρό των εταίρων της και θα τιμά τις συμφωνίες που θα έχει κάνει και τις ευθύνες της. Έτσι ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν περισσότερα για την ασφάλεια και την αμυνά του. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο ρόλο τη Στρατιωτικής Επιτροπής είναι ρόλο ε, δημόσια διπλωματία. Ε, θεωρώ ότι μια τέτοια αναβάθμιση θα βοηθήσει και τη Στρατιωτική Επιτροπή να μπει σε συζητήσει με το Βιετνάμ, ε, τη Μιανμάρα, το Πακιστάν και αργότερα ενδεχομένω με την Ινδία. Αυτή η προσπάθεια σε συνδυασμό με τη συμμετοχή αξιωματούχων ε, σε διάφορα μαθήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις θα αυξήσει την αναγνώριση του στρατιωτικού σκέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό στα μέλη της Επιτρόπης αυτής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα τις στρατιωτικές της ε, δυνάμεις. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει να βρει εταίρους που θα συμβάλλουν στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της. Κατανοώ το ότι το να έχουμε εταίρους στις αποστολές και τις επιχειρήσεις μας δεν αντιμετωπίζει απλά τα πρακτικά προβλήματα έλλειψης προσωπικού και ικανοτήτων, αλλά βελτιώνει και την εικόνα που δίνουμε στον κόσμο, ε, όπως περιγράφεται στην παγκόσμια στρατηγική και στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλάμε για πολλούς εταίρους που συνενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώ εγώ τις καλές προσωπικές σχέσεις που έχω δημιουργήσει στα ε, δεκαετή μου ε, καριέρα ε, ως επιτελάρχη ώστε να ζητήσω από τη Βοσνία Ζεγοβίνη και άλλους να συμμετέχουν στις δικές μας αποστολές ως εταίροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποφάσισαν από κοινού να ενισχύσουν την συνεργασία τους. Όπως αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη του Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή συμβάλλει με τη διοργάνωση άτυπων και τυπικών συναντήσεων του ΝΑΤΟ στο κατάλληλο επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι πρόεδροι των αντίστοιχων επιτροπών καλούνται να συμμετέχουν στις ε, συνεδριάσεις ε, των επιταλαρχών ε, του άλλου οργανισμού. Μια άλλη προσωπική μου άποψη που προσπαθώ να υλοποιήσω αφορά τη σύνθεση του γραφείου μου. Το προσωπικό μου, Είναι κατάλληλο, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη ε, στο προσωπικό μου, όχι να έχω μόνο ε, προσωπικό από τη δική μου χώρα, να ε, υπάρχει εκπροσώπηση από όλε τι στρατιωτικέ δυνάμει. Και σήμερα το γραφείο μου αποτελείται από αξιωματούχου από 14 διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα κλείσω εδώ κυρίε και κύριοι και περιμένω τι ερωτήσει σα. Πριν από αυτό θα ήθελα να αναφέρω επί τη ευκαιρία ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν λάβει χώρα ρηξικέλευτε αλλαγέ ε, στον τομέα τη άμυνα και της ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με περηφάνεια πρέπει να πω ότι η Στρατιωτική Επιτροπή, εγώ και το προσωπικό μου, έχουμε παίξει έναν μετριοπαθή αλλά πρέπει να πω σημαντικό ρόλο ώστε να εκπληρώσουμε το όραμα της παγκόσμιας στρατηγικής και να ενισχύσουμε την Ευρώπη. Αλλά για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα απαιτείται πάθος, δέσμευση και ε, ε, επιμονή. Έτσι λοιπόν στους 10 μήνες που απομένουν μπροστά μου ως Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής θα συνεχίσω να αφιερώνω όλη μου την ενέργεια σε αυτή την Επιτροπή και στην εκπροσώπηση των κρατών μελών και των προτεραιοτήτων. Σας ευχαριστώ. Sir, thank you very much for the... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ, για αυτήν την πολύ σημαντική συμβολή σας. Ένα μέλος της Επιτροπής μας έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Γκάλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Στρατηγέ, σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή μας. Να σα ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά και για τους επόμενους δέκα μήνες βεβαίω. Αλλά όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε σε πολλές ε, πρακτικές αλλά και πολιτικές πλευρές των ζητημάτων που σας απασχολούν καθώς και οι επιθυμίες που εκφράσατε όσον αφορά την πολιτική βούληση ε, την χάνουν και της δική μου ε, συμφωνίας. Προς το τέλος της ομιλίας σας αναφερθήκατε σε κάποιες καινοτομίες στον ε, τομέα της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Είναι και αυτό μια έκφραση πολιτικής βούλασης. Ε, χωρίς πολιτική βούληση δεν θα είχαμε καταλήξει στην ΠΕΣΚΟ άλλωστε. Επομένως το ζητούμενο τώρα είναι να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ορατή, να γίνει ορατή και η προστιθέμενη αξία αυτών των αποφάσεων. Και από τη σκοπιά αυτή θα έλεγα ότι τα έργα και τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ε, θα ήθελα να μου πείτε τι ελλείψεις έχουν μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σας κατά τη γνώμη μου τα, τα προγράμματα αυτά δεν είναι τόσο φιλόδοξα. Θα μπορούσαν ενδεχομένω να είχαν υλοποιηθεί και χωρίς την ΠΕΣΚΟ δηλαδή. Από αυτή την άποψη έχετε κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσαν να καταρτιστούν πιο φιλόδοξα σχέδια. Ίσως ε, η, η οικοδόμηση και η δημιουργία ενός γενικού επιτελείου το οποίο θα, θα είναι άξιο του ονόματός του θα μπορούσε να αναλυφθεί στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ. Επίσης, πρέπει να δείξουμε στην παγκόσμια κοινότητα ότι μπορούμε να κάνουμε, ότι έχουμε πράγματι μια σκληρή στρατιωτική δύναμη, hard power όπως είπατε και εσείς, ε, και να μπορεί να το επιδείξει αυτό για τις μάχημες ομάδες. Ορθώς είπατε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αφενός γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση, αφετέρου γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Συζητούμε εδώ και χρόνια ε, για την ε, διεύρυνση του μηχανισμού Αθηνά. Μήπως μια βαθμιαία προσέγγιση θα περιλάμβανε το εξής. Ναι, μάχημες ομάδες όποτε ε, τίθενται ε, σε εφαρμογή και σε επιχείρηση πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως και ενδεχομένως και από ξεχωριστό κονδύλιο. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει κατά τη γνώμη σας ένα πρώτο βήμα. και να χρηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο και το προσωπικό αλλά και ο υλικός εξοπλισμός που χρειάζεται για την ανάπτυξη τέτοιων ε, μονάδων. Και τέλος, έχετε πρακτική εμπειρία γνωρίζετε ποιες είναι οι αποστολές μας, οι επιχειρήσεις μας. Γνωρίζετε ποιες είναι οι ανάγκες και έχουμε και αυτόν τον ε, το μηχανισμό CARD όπου όλοι οι φορείς ε, σχεδιασμού υποβάλλουν τις δικές τους πληροφορίες, τι χρειάζονται, τι απαιτείται. Ζητούμενο είναι να βρεθεί και ένας τρόπος ε, συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών. Αυτός, είναι, αυτό, αυτό, αυτό αυτός ο μηχανισμός, ο, ο CARD, να υπάρχει, να υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός και μια γενι, γενικός και, κοινός, και κοινή ανάπτυξη επιχειρήσεων. Ο κύριος Στατίνα. Děkuji vám za slovo, paní Λοιπόν. Ευχαριστώ που, που μου έδωσε το λόγο, Πρόεδρε. Στρατηγία, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Επ' θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις δράσεις σας ε, για την επιχείρηση Σοφία στο Τσάντ στη Λιβύη και στη Λιβύη και στη Σομαλία φυσικά. Όμως, θα ήθελα να σας πω ότι ο πόλεμος ο οποίος είναι πραγματικά στην αυλή μας, στη γειτονιά μας, δίπλα μας, είναι στην Ουκρανία. Λίγες ώρες με το αυτοκίνητο απέχει αυτή η χώρα. Και ξέρουμε ότι μια πολιτική λύση πόρο απέχει από το να βρεθεί. Η συμφωνία Μίνσκ δεν σταμάτησε τις μάχες και το χύσιμο αίματος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, στρατηγέ, ως ε, αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, πώς θα λύνατε εσείς την Ουκρανική σύγκρουση, την Ουκρανική σύραξη, δεδομένου του ότι ε, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο πριν από λίγες μέρες είπε ότι κάνει τώρα επιχειρήσεις αντιτρομοκρατικές. Καταπολεμάει την εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη χώρα. Στρατιωτικός πώς, πώς θα επιλύεται αυτή την κατάσταση. Αν μπορούσατε να κλείσετε τα, τα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Στατίνα. Ε, συμφωνώ και εγώ με αυτό το ερώτημα που υποβλήθηκε για την Ουκρανία και εγώ θα υποβάλω και ένα επιπρόσθετο ερώτημα. Ο κύριος Κάρβε που είναι ο συντονιστής τώρα. Ε, πώς έχει λυθεί το θέμα των, ε, μονα, ε, μονάδων, ε, των μάχημων μονάδων μετά το θέμα του Brexit. Γιατί συμμετείχανε, συμμετείχε το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτές τις μονάδες. Επίσης, θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια σκέψη για τη Σομαλία. Τι σκέψεις κάνετε για το πώς θα καλυφθεί το κενό που υπάρχει στη Σομαλία. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μια μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή αυτή. Ε, ε, Ευχαριστώ, στρατηγέ. Κύριο Ομολογώ ότι μου άρεσε πολύ η παρουσίασή σας. Έχω την αίσθηση ότι είστε ένας εξαιρετικός επικεφαλής ε, των στρατιωτικών, των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ε, ευχή έργο να έχουμε αντίστοιχους ηγέτες και στο πολιτικό επίπεδο. Η νέα πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφηθεί καταδεικνύει ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Με βάση, με βάση όμως τη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε, είμαστε αντιμέτωποι και με μια σειρά νέα στοιχεία. Πολλοί παρατηρητές έχουν την αίσθηση ότι οι διακηρύξεις αυτές περισσότερο στα λόγια μένουν παρά υλοποιούνται. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις λοιπόν. Η Στρατητική Επιτροπή ε, είναι αρμόδια να καταρτίζει τον κατάλογο απαιτήσεων. Μιλούμε για μια κοινή πολιτική. Και βλέπουμε ότι ο κατάλογος αυτός απαιτήσεων, παρότι καταρτίζεται, ε, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένους ορισμούς ακόμη. Είναι νέο καθήκον αυτό που εκκρεμεί ακόμα. Και δεύτερον, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, που έχει ως ρόλο να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, ώστε να έχουμε κοινή έρευνα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού του οργανισμού, πώς θα την αξιολογήσετε, ε, ποιες, ποιους στρατιωτικούς πόρους θα, θα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε ακριβώς την αποτελεσματικότητα αυτή. Κύριος Φρόιντ, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον στρατηγό για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ενωσιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα ε, στο θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη και διορθώστε με αν κάνω, ε, αν λάθος είναι μια χώρα όπου η κατάσταση που υπάρχει σήμερα ε, υπάρχει εκεί εδώ και 10 χρόνια. Και αναρωτιέμαι δεδομένου ότι τμήμα της αποστολής αυτής και καθήκον της είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων του Βοσνιακού στρατού, γιατί χρειάστηκαν περισσότερα από 10 χρόνια, ώστε να καταστεί έτοιμη, ε, έτοιμες οι να καταστούν έτοιμε οι ένοπλες δυνάμει προκειμένου να αναλάβουν το έργο το οποίο υποτίθεται ότι ε, καλούνται να εκπληρώσουν. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα αυτή γιατί δεν λειτουργήσε το πρόγραμμά μας μέχρι στιγμής. Σχετίζεται αυτό με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Σχετίζεται μήπως ε, με το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί γιατί αυτό παρέχει σταθερότητα και στο στρατό και στην ίδια τη χώρα ή μήπως έχετε παρετηθεί από το καθήκον της ε, ανάπτυξης ικανοτήτων. Πείτε μου εσείς ε, ποιο πιστεύετε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρόβλημα στη Βοσνία. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος, στρατηγέ. Για την επίσκεψή σας στο Βιετνάμ, θα ήθελα να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Νοτιοανατολική Ασία, δεδομένων και των κινήσεων ε, στρατιωτικής ανάπτυξης της Κίνας και της κινήσεις ελευθερίας πλοήγησης ε, στην περιοχή, αλλά και την συμμετοχή και την ε, εμπλοκή άλλων εμπλεκομένων χωρών της συγκεκριμένης περιφέρειας. Και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εκεί. Επίσης, ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία ποια είναι η κατάσταση της, ε, των συμμαχικών δυνάμεων που δρούν εκεί, αλλά και πιθανές εξελίξεις εν ώψη της τουρκικής επίθεσης. Αυτά. Ολοκληρώσαμε τις ε, ερωτήσεις. Ε, Στρατηγία, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ άριθμες ερωτήσεις. Μεγάλη σημασία Πρόκειται για τα στατικά στοιχεία που παρέλειψα να σας παρουσιάσω, γιατί δεν είχα αρκετό χρόνο να μπω και σε αυτά. Ας ξεκινήσω από τα project Το θέμα της διαρθωμένης συνεργασίας, του μόνιμης διαρθωμένη συνεργασίας, ε, κινήθηκε γοργά. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο χρονισμό, το χρονοδιάγραμμα δεν είναι κλασικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινείται μέσα σε λίγου μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο σημαντικά project όπω αυτό ε, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και όλοι μα ε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Για την υπογραφή της ΠΕΣΚΟ σε υψηλότατο επίπεδο σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο αποφασίστηκε να υπάρξουν διάφορα αρχικά project. Μια πρώτη δέσμη project που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πάρα αυτά. Άλλα project, άλλα έργα, τα οποία απαιτούσαν υποδομή ή, εν πάση περιπτώσει, πολλές πολιτικές συζητήσεις. Πέρασαν στη δεύτερη δέσμη project, γιατί χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν. Όλα αυτά λοιπόν τα project είναι αυτά που ξεκινήσαμε ήδη να υλοποιούμε και οι χώρες δέχτηκαν αυτές τις ε, καθοδηγήσεις, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και πιστεύω ότι πριν από το τέλος του 18 θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Υπάρχουν ε, πολλά πράγματα που είναι αναγκαία. Υπάρχει ένα project ε, της Γερμανίας για ένα σώμα στρατού που θα ασχοληθεί με θέματα διαχείρισης κρίσεων και καλύπτει μία γκάμα διαφόρων δυνάμεων. Υπάρχουν και άλλα project πολύ σημαντικά και αν υλοποιηθούν όπως αναμένουμε, αν συμφωνηθούν από τα κράτη-μέλη, τότε θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες, θα έχουμε στρατιωτική κινητικότητα, που είναι ένα τεράστιο θέμα. Και άλλες οργανώσεις ε, δουλεύουν επί χρόνια για να την υλοποιήσουν και να την πετύχουν. Είναι ο βασικός λόγος για τις επιλογές που κάναμε για την πρώτη δέσμη προγραμμάτων. Θα ξεκινήσουμε την επίσημη αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Και για κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη, τα ηγετικά κράτη-μέλη, ε, κάνουν ήδη κινήσεις και ασχολούνται ήδη με το θέμα. Τώρα για τις α, μάχημες μονάδες. Όταν ξεκινήσαμε να δημιουργούμε αυτό τον ε, στρατιωτικό βραχίωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιγράψαμε τον ΝΑΤΟ. Ε, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση. Γιατί όπου το κόστος, ας πούμε, αντιμετωπίζεται εκεί που γεννάτε. Είναι λογικό για τον ΝΑΤΟ. Είναι μια μεγάλη δύναμη, ένα μεγάλος οργανισμός. Όταν έχουμε, ας πούμε, ένα καθολικό πόλεμο, ε, έναν πυρηνικό πόλεμο, <laughs> τότε δεν αρχίζουμε ερωτήσεις του ποιος πληρώνει τι. Αλλά εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοιου τους πολέμους. Ε, έχουμε να κάνουμε με την αντιμετώπιση κρίσεων. Και μία κυβέρνηση, ας πούμε, που ξοδεύει χρήματα για να επιληθεί μια κρίση σε άλλα τμήματα του πλανήτη, για, για κρίσεις που δεν τις αφορούν άμεσα, έτσι. Δεν συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούν να δικαιολογήσουν στους πολίτες το γιατί δαπανούν αυτά τα χρήματα. Γιατί για τους επόμενους έξι μήνες θα στείλουμε ας πούμε, μάχινες μονάδες στη χώρα Χ, ας πούμε, και αυτό μας κοστίζει ας πούμε 100.000 ευρώ. Και προσπαθούν να το αποφύγουν αυτά τα κράτη-μέλη, γιατί το κόστος είναι υψηλό. Η άμυνα είναι πολύ ακριβώς σπόρο. Το να στέλνεις μια φρεγάδα, ε, φρεγάτα συγγνώμη, κάπου στον Ινδικό ωκεανό για να υποστηρίξει την επιχείρηση Αταλάντα, σου κοστίζει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια το μήνα. Έχεις τα άτομα αυτά για 4, 4 μήνες εκεί θέλεις 12 εκατομμύρια. Εντάξει. Το να έχει, ας πούμε επιπλέον έξοδα κάπου μέσα στον, στη χρονιά σου α πούμε σου δημιουργεί προβλήματα και τρύπε στον προπολογισμό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν και άλλου μηχανισμού. Και η Αθήνα δεν είναι αρκετή ικανή επιχείρηση για μας. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι στις συνθήκες δεν προβλέπεται να δώσει κομισιόν λεφτά σε, στα, για στρατιωτικά θέματα. Όταν περνά μέσω της κομισιόν δεν γίνεται τίποτα. Εν τη περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και αν δεν τα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όπως πρέπει τις μάχημες αυτές μονάδες εκεί που πρέπει. Για ε, το θέμα του ΚΑΡΝΤΑ, την ολοκλήρωση της ετήσιας ανάλυσης για την άμυνα. Εμείς έχουμε το μηχανισμό για την ανάπτυξη στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων για την ΚΠΑ. Έχουμε τον κατάλογο απαιτήσεων Όλα αυτά τα συντάσσουν οι εμπειρογνώμονες της Στρατιωτικής Επιτροπής και δίδονται στην ε, EDA και να συνταχθεί ε, το σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων. Είμαστε σε στενή επαφή, παρακολουθούμε και εμείς τη διαδικασία και το κάνουμε αυτό για να εγγυηθούμε ότι όσοι ασχολούνται με τις επιχειρήσεις θα αποφασίσουν για τις ανάγκες και δεν θα αποφασίσει η αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε εκεί και είμαστε σε κάθε βήμα. Γιατί όσοι ασχολούνται με τις διάφορες επιχειρήσεις ε, από τις διάφορες χώρες το, και από τις 28 χώρες δηλαδή, είναι παρόντες ούτω ώστε να μας πούν τι χρειάζονται. Και δεν αφήνουμε ας πούμε την αμυντική βιομηχανία, τον, αμυντικό, τομέα να μας πει τι χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι κάνουμε μια καλή και γρήγορη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Πρέπει να έχει εμπειρογνώμονες. Η δουλειά είναι πολύ λεπτομερής, αλλά και εμείς κινούμαστε γρήγορα, γιατί χρειαζόμαστε την ΚΠΑ και όλη αυτή η προσπάθεια θα βοηθήσει το CARD. Ε, είναι μία από, ένα από τα σκέλη που κινούνται ταχαίως. Θα είναι σε δοκιμαστική φάση πολύ γρήγορα και όπως και η ΠΕΣΚΟ πάει πολύ καλά. Και η ΠΕΣΚΟ και η ΚΑΡΤ πάνε μια χαρά. Τώρα για την Ουκρανία. Το στρατιωτικό σκέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, οι στρατιωτικές δυνάμεις τη Ευρωπαϊκής Ένωση, της Ευρωπαϊκής δεν ασχολούνται, δεν έχουν παρέμβει στην Ουκρανία καθόλου. Αυτό που κάνουμε για να υποστηρίξουμε του εταίρου μα στην Ουκρανία είναι ότι προσκαλούμε τον αρχηγό Γεθά στις ε, συνεδριάσεις μας για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Ε, δεν υπάρχει εντολή για αποστολή, δεν υπάρχει αποστολή, δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει τίποτα στην Ουκρανία. Υπάρχει μια μη στρατιωτική αποστολή εκεί, στην Ουκρανία, είναι κάτι άλλο, ένα άλλο τομέα. Δυστυχώ δεν μπορώ να σα πω τίποτα για αυτή την αποστολή. Τώρα, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά πώς θα επέλεια το πρόβλημα της Ουκρανίας, να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι με την προστασία της Ευρώπης και όχι με την άμυνα της Ευρώπης. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε προβλήματα με, αυτή, με όλη την, αυτή την ανάπτυξη αμυντικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι διευκρινίσαμε στο ΝΑΤΟ ότι η άμυνα της Ευρώπης είναι, ανήκει στο ΝΑΤΟ και ασχολείται με αυτό, ενώ η προστασία της Ευρώπης είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς με πολύ δραστήριο τρόπο ασχολούμαστε γι' αυτό. Με, τον, με την μετανάστευση τον ε, έλεγχο των συνόρων, δηλαδή, κατά πολέμηση τρομοκρατίας κτλ. Επομένως έχουμε κάνει αυτή τη διαίρεση και κρατάμε αυτές τις αρμοδιότητες που μπορούμε. Λόγω αυτού δεν μπορώ να σας πω κάτι για την Ουκρανία, ε, λυπάμαι παρότι είναι μεγάλο, πηχαίο τίτλος, εγώ δεν είμαι ε, αρχηγός ΓΕΘΑ στην πραγματικότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει αρχηγός ΓΕΘΑ. Είμαι επικεφαλής της Στρατιωτικής ε, Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ε, μία θμίδα κάτω από το Θεό. Εγώ είμαι ένας απλός πρόεδρος. Και αυτό είναι το σημαντικό ε, που υπάρχει στην οργάνωσή μας και θα πρέπει να είμαστε ε, περήφανοι γι' αυτό. Είμαι, εγώ είμαι εκλεγμένο. Είμαι ο μόνος εκλεγμένος, ας πούμε, ε, στρατιωτικός. Συνήθως διορίζονται στις, ε, στους στρατιωτικούς σχηματισμούς οι άνθρωποι. Εμείς εκλέξαμε τον πρόεδρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δίνει επιπλέον ε, ισχύει και εξουσία σε αυτό το άτομο. Γιατί εκπροσωπεί πραγματικά τα 28 κράτη-μέλη, αλλά δεν διοικεί στρατεύματα. Δεν διοικεί στρατεύματα. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω για την Ουκρανία είναι ότι πάντα προσπαθούμε να γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση στη χώρα, αλλά μια και δεν υπάρχουν αποστολές, μια και δεν υπάρχει πολιτική βούληση για οποιαδήποτε εμπλοκή συμμετοχή δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Για τις μάχημες μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν μια πολύ σημαντική συνεισφορά στρατιωτικά του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή. Δυστυχώς θα αντικατασταθούν. Όλες οι μάχημες μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου στις επιχειρήσεις μας, το OHQ, για την επιχείρηση Αταλάντα και το Northwood, όλε αυτέ οι μονάδε θα αντικατασταθούν, μια και το Ηνωμένο Βασίλειο Δυστυχώ αποφάσισε να φύγει, Δυστυχώ για μα. Θα βρούμε λύσει. Υπάρχουν και άλλε μονάδε, μάχημε μονάδες από άλλε χώρε. Πρέπει να σα πω ότι το, η δυσκολία είναι ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ποιότητα των Βρετανών συναδέλφων που είναι ικανότατοι, τα στρατεύματα αυτά είναι υψηλού ποιοτικού επίπεδου, πολύ επαγγελματικά, έχουν μεγάλη πείρα, ε, φοβερή παράδοση. Ένας ε, πολύ, πολύ καλό στρατός παραδοσιακά είναι ο Βρετανικός. Αυτό που λέω στους φίλους μας, όταν μας ρωτάνε αυτές τις ερωτήσεις, είναι ότι τι να σας πω, εμείς δεν αποφασίσαμε να φύγουμε. Οι Βρετανοί θα αποφάσανε οι ίδιοι να φύγουν και εμείς θα βρούμε απλώς λύση για να τους αντακαταστήσουμε. Είναι θλιβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα στρατηγέ, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Απλά ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς έχουμε άλλα δύο λεπτά μόνο. Εντάξει, κανένα πρόβλημα δεν έχω αυτό. Για το ETA και τον οργανισμό δεν μπορώ να σας πω ε, ακόμα κάτι για την αποτελεσματικότητα. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνεται στην κυρία Μογκερίνη. Εκείνη είναι υπεύθυνη. Δυστυχώ επίση δεν μπορώ να σα πω τίποτα για την κατάσταση στη Δεν παρεμβαίνουμε εκεί. Ούτε μπορώ να σα πω κάτι για την ε, ε, τουρκική επιχείρηση, αν και είναι προφανέ το τι κάνουν. Ε, επίσκεψη στο Βιετνάμ. ναι, προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε το Βιετνάμ. Η θέση μας και την οποία τους δηλώσαμε και την έχουμε ε, πει και στους Κινέζους είναι ότι θέλουμε ειρηνική λύση στην Νότια Κινέζικη θάλασσα βάσει των ε, αποφάσεων του ΙΕ και βάσει του δικαίου της θάλασσας. Τη σύμβαση για τη θάλασσα. Την Ούγκλος. Αυτό λοιπόν κάνουμε ε, με την UNCLOS που είναι το βασικό μας εργαλείο. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν. Τα πολιτικά προβλήματα έτσι και δεν επιλύονται στρατιωτικά. Δεν είναι ανέφικτο και να θέλει κανείς. Και αυτό κηρύσουμε. Αν έχετε πολιτικά προβλήματα, πρέπει πολιτικά να τα επιλύσετε. Μην προσπαθείτε να βρείτε στρατιωτικέ λύσεις σε πολιτικά προβλήματα. Για τη Βοσνία. Ναι, χρειάστηκαν 10 χρόνια. Έχουν πλέον ε, ένοπλες δυνάμεις, στρατό, αλλά μην ξεχνάτε ότι η αφοσίωση και η προσήλωση των ε, πολιτών της χώρας αυτής ανήκει στις κοινότητες του καθενός. Δεν ξέρουμε λοιπόν σε ποιο βαθμό ε, θα διαφυλαχθεί η αμεροληψία αυτού του στρατού. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο τους εκπαιδεύουμε, αλλά ξέρετε ότι σε όλες αυτές τις χώρες η οικογένεια, η τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει κανείς είναι πολύ ισχυρό μέγεθος στη ζωή ενός ανθρώπου αφοσίωσή τους λοιπόν και η προσήλωση των ανθρώπων στην Βοσνία Ρεζεγοβίνη κατά κύριο λόγο ανήκει στην κοινότητα στην οποία ανήκει ο καθένας. Οι στρατιωτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά γνωρίζετε κι εσείς ότι οι πολιτικές ηγεσίες είναι αυτές που δεν συνεννοούνται και δεν συνεργάζονται καλά και εδώ πρέπει βεβαίως να βρεθεί λύση, αλλά είναι πολιτικό και αυτό το θέμα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι προσπαθούμε να, να βάλουμε τη χώρα αυτή να λειτουργήσει στη βάση, με βάση τη συμφωνία του Dayton. Η συμφωνία του Dayton ήταν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μετά τον πόλεμο. Η χώρα αυτή πλέον έχει σύνταγμα και πρέπει να το εμπλουτίσει αυτό το σύνταγμα. Να το συμπληρώσει με συγκεκριμένες ε, συνταγματικές διατάξεις και να ξεφύγει η χώρα από τη συμφωνία του Ντέιτον, η οποία ήταν χρήσιμη και καλή όταν συνήφθη για να σταματήσει η αιματοχυσία. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Γι' αυτό και χρειάζεται οι κύριες προσπάθειές μας να κατευθυνθούν στο να επαναδιευθετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτό είναι το βασικό ε, καθήκον και νομίζω ότι μέχρι, μέχρι τούδε πολιτικές πρωτοβουλίες δεν κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ στρατηγέ για την παρουσία σας και για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας και η συζήτησή, σας, η συζήτησή μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία βεβαίως και για τους επόμενους δέκα μήνες αλλά και για την για το επόμενο διάστημα μετά την ε, ολοκλήρωση της θητείας σας και ε, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την ε, επιτυχή έκβαση των στρατηγικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να χειροκροτήσουμε τον στρατηγό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ παραμείνετε. Έχουμε το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα με έναν σημαντικό ομιλητή στην ημερήσια διάταξη.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 Παρακαλώ καθίστε. Ξεκινάμε αμέσως με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε τον διακεκριμένο προσκεκλημένο μας, τον αντιστράτηγο αποστρατεία του Βουλγαρικού στρατού, αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της χώρας που αυτή τη στιγμή για το επόμενο εξάμενο προεδρεύει ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη μου τιμή λοιπόν και ευχαρίστηση καλωσορίζω τον ε, ε, στρατηγό Ατάνας Ζαπριάνοφ στην ε, συνάντηση της ΣΕΝΤΕ. Χαίρομαστε ιδιαίτερα που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση ενημέρωσης και επαφή με εσά, κύριε Αντιστράτη, και σα δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσετε τι απόψει για τι εξελίξει ε, ε, στην ε, κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και τι προτεραιότητε τη Βουλγαρική Προεδρία. Εγώ είμαι Πολωνή, οπότε κάθε προεδρία της δικής μου περιφέρειας είναι πολύ σημαντική, και την υποστηρίζουμε. Συζητήσαμε εκτενώς τα ζητήματα της ασφάλειας ε, στην περιοχή του Εύξενου Πόντου καθώς ε, και την ε, ασφάλεια και τα θέματα άμυνας στα Δυτικά Βαλκάνια. Σίγουρα αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Έχετε λοιπόν το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε με μεγάλη μου χαρά και τιμή παίρνω το λόγο μπροστά σε τόσο έμπειρο ακροατήριο. Τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, που εμπλέκεται άμεσα στα θέματα ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στον τομέα της άμυνας. Έχουμε τέσσερις προτεραιότητες ως Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοχή και συνέχεια με τις υπόλοιπες προτεραιότητες ε, ε, του Τρίου Προεδριών και ταυτόχρονα είναι προτεραιότητες που αντιστοιχούν στις δικές μας ιδέες. Οι πρώτες μας προτεραιότητες και η ενεργός μας ε, υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Παγκόσμιας Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας και της Ασφάλεια, συνεχίζουμε όλες τι προσπάθειες για να αναπτύξουμε πρωτοβουλίε που προκύπτουν από την παγκόσμια στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Από αυτή την άποψη η Βουλγαρία συμμετέχει στην ανάπτυξη της ε, μόνιμης δομής στον τομέα της ε, Άμυνα και στην επιτυχή έναρξη των τεσσάρων ε, έργων που είναι υψηλού πολιτικού και δημοσίου ενδιαφέροντο. Μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μα. είναι η προσαρμογή του κανονισμού περί δημιουργίας ε, ενός ευρωπαϊκού ε, προγράμματος ε, ευρωπαϊκής αμυντικής μηχανίας. Είναι σημαντικό για την δημιουργία δυνατοτήτων στρατιωτικών και για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συμμετοχών χωρών με τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχείρησεων σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των χρηματοδοτήσεων. Έχει υψηλή προτεραιότητα αυτό το ζήτημα για την προεδρία μας. Θα το αναλύσω λιγότερα, λιγο, περισσότερο αργότερα. Η δεύτερη μας προτεραιότητα είναι η υποστήριξη για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Προεδρία. Θέλουμε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανάπτυξη προτεραιοτήτων και το σχετικό σχέδιο, η ανάπτυξη δυνατοτήτων και το σχετικό σχέδιο και να συμμετέχουμε στη συντονισμένη αναθεώρηση της άμυνας. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικός παραγόντας η γεωπολιτική ασφάλεια στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο η τρίτη μας προτεραιότητα που είναι η σταθεροποίηση της ασφάλειας ε, στα Βαλκάνια είναι σημαντική. Όσον αφορά την άλλη ε, προτεραιότητα αυτή, η πρωτοβουλία, την ε, ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, εστιαζόμαστε στην ασφάλειά τους. Αυτό θα ξεκινήσει η Βουλγαρική προεδρία και μετά η αυστριακή και οι ρουμάνοι συνάδελφοι θα την συνεχίσουν. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία να επιτύχουμε κάποια επικοδομητικά αποτελέσματα προς όφελος της ευρωπαϊκής ε, ασφάλειας και συνεργασίας για να αποφύγουμε περί επανάληψη εργασιών ε, χρειάζεται συνοχή στις πολιτικές ε, στον τομέα της άμυνας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο η τέταρτη μας προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δυνάμει τη ε, διακήρυξη της Βασοβίας. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο ε, τον αποφεύγουμε οποιοδήποτε διπλασιασμό των προσπαθειών μεταξύ των δύο οργανισμών είναι μια άριστη ευκαιρία εξοικονόμησης χρημάτων των φορολογουμένων τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο μας για το νέα δέσμη μέτρων για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υλοποιείται υπό το πνεύμα της διακήρυξης τη Βαρσοβίας. Θα υπογραμμίσουμε την πρακτική συνεργασία στον τομέα για να λειτουργήσουν όλα αυτά και για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεται να διοργανώσει 28 ε, συναντήσεις ε, 12 στις Βρυξέλλες και 16 στην Βουλγαρία. Για να σας αναφέρω τις σημαντικότερες άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας και σεμινάριο υψηλού επίπεδου για τις ευκαιρίες ε, οικοδόμησης και υποστήριξη δυνατοτήτων στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, σε ε, διάσκεψη υψηλού επίπεδου ε, για την έρευνα και την τεχνολογία και τη βιομηχανική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και για τι καινοτομίε στον χώρο. Υπάρχουν και κάποιες μακροχρόνιες προκλήσεις και ευκαιρίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά όσον αφορά την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Η άμυνα και η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Είναι κάτι επιβαλλόμενο. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα βρίσκονται στη θέση του οδηγού καθώς θα καθορίζουν και θα υλοποιούν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι πρωτοβουλίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή καταδεικνύουν σαφώς ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη ε, αναλάβει αυτό το ρόλο. Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί το πόσο γρήγορα θέλουν τα κράτη-μέλη να οικοδομήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας και μετά να απαντήσουν και ερωτήματα όπως σε ποιο βαθμό επιθυμούν να υπάρχει πρόβλεψη αντί για αντίδραση ε, σε στρατηγικό πλαίσιο σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί ευρωπαϊκή ευθύνη. Η Βουλγαρία αναγνωρίζει ότι μία από τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στην οικοδόμηση μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση είναι ο κίνδυνο οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση εθνικιστική ε, Ευρώπη. Ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τους βασικούς, τις βασικές πηγές που τροφοδοτούν ε, το λαϊκισμό, τον εθνικισμό σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Τέσσερις ε, πρωτοβουλίες πολιτικής που προωθήθηκαν κατά το περασμένο έτος αποτελούν σίγουρα ευκαιρίες θετικές. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν αμοιβαία και να ενισχύσουν τις ε, δομές σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανέφερε και ο στρατηγός ο κ. Κωνσταράκος. Στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε διαδικασίες τακτικής αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Άμυνας και του συντονισμένης αναθεώρησης της άμυνας να ξεκινήσουμε μόνιμη στρατιωτική συνεργασία, ε, τη μόνιμη δομή συνεργασίας για τις χώρες που είναι έτοιμες να επενδύσουν περισσότερο, να συνεργαστούμε για πιο φιλόδοξα ε, έργα δημιουργίας ικανοτήτων ε, και να συμμετέχουμε με δυνάμεις σε διάφορες δυνάμεις. Και ξεκινώντας το Ταμείο Άμυνα, το οποίο θα υποστηρίζει την έρευνα για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Θεωρούμε ότι η εξωτερική και εσωτερική ε, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ε, την κατάσταση μεταξύ κρατών μελών ε, και να καταλάβουμε και ποιες δράσεις απαιτούνται για το μέλλον. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να εστιαστούμε στην καθιέρωση φιλόδοξης ε, συνεργασίας ε, στο πλαίσιο μιας μόνιμης δομής ε, χωρί αποκλεισμού και με τη χρήση των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί κατά πολλούς τρόπους από την διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών κινήτρων ώστε να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποια βασικά project που θα καλύπτουν την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τις επιχειρήσεις και τις δύο διαστάσεις αυτές μα ενθαρρύνει η έναρξη των πρώτων λεπτά έργων στον τομέα της ε, ΠΕΣΚΟ. Η Βουλγαρία θα συμμετέχει σε τρία από αυτά και θα είναι ε, παρατηρητής σε κάποια άλλα. Η Βουλγαρία αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να συντονίσουμε την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού άμυνας ώστε να ενισχύεται η αποκρισή μας, να ενισχύονται οι δυνατότητες σχεδιασμού και να αναθεωρούνται οι κανόνες ε, για το κοινό ε, θεμέλιο των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. thank you very much. Ευχαριστώ Υπουργέ για την ολοκληρωμένη εισήγησή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της Επιτροπής μας. Κύριε Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω Υπουργέ, σας και την ε, το επιτελείο σας στην υποεπιτροπή μας. Κάθε ευχή για όλο το 2018 και ιδίως για το πρώτο εξάμεινο αυτού, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που αναλαμβάνετε την Προεδρία του Συμβουλίου, μια νέα εμπειρία για σας. Έχω μιλήσει όμως και με άλλες χώρες που ανέλαβαν για πρώτη φορά στο παρελθόν την Προεδρία και με επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ζωή και μετά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ε, έχουμε ενεργοποιήσει πρόσφατα την ΠΕΣΚΟ και όλα τα παρατήματα που την συνοδεύουν. Όλα πλέον βρίσκονται σε πλήρη ε, επιχειρησιακή ανάπτυξη και εσείς ε, έχετε τον άχαρο ρόλο να δείτε πώς όλα αυτά θα τελικά θα συνδυαστούν. Τα ταμεία, τα, τα προγράμματα, η χρηματοδότηση, οργανισμός, όλα αυτά πλέον ε, έχουν αποφασιστεί, έχουν τεθεί επιτάπητος και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει ένας συντονισμός. Πρώτα απ' όλα βεβαίως είναι το CARD, η αναθεώρηση δηλαδή, αυτό για να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε και τι χρειαζόμαστε, ποιες είναι οι ανάγκες. Πρέπει επίσης να προσδιοριστούν και άλλα ε, προγράμματα, έργα, στον τομέα της έρευνας, στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων, και βεβαίως υπάρχει και η δημοσιονομική διαδικασία ε, που προβλέπει την συνεισφορά ε, των κρατών μελών συν 20% από την Κομισιόν. Έχετε λοιπόν κάποια επισκόπηση, κάποια εποπτεία για το πώς τελικά θα γίνει αυτός ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων, σωμάτων ε, Βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ. Ποια είναι η θέση του, του Συμβουλίου, Ιδίω και ως προς την ε, συνεργασία, της με την, ε, συνεργασία του με την Κομισιόν, καθώς ε, για πρώτη φορά εμπλέκεται σε ζητήματα άμυνας η, η Κομισιόν. Αυτό. ένα δεύτερο ερώτημα. η χώρα σας βρέχεται από τον Εύξηνο Πόντο, ε, από τον οποίο βρέχεται και η Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή επιτίθεται στη Συρία. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ να αναλαμβάνει τέτοιου είδους ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και κάποια άλλη άποψη. Ίσως εσείς εκτιμάτε διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, η Ρωσία ε, μέσω της ε, προσάρτησης της Κρυμαίας επίσης ε, ήρθε πιο κοντά στη Μαύρη Θάλασσα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, εμείς ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς στο Συμβούλιο τι κάνετε στην... και σε συνεργασία και με τη Ρουμανία πώς συνεργάζεστε με όλους τους εταίρους για να παρακολουθείτε πιο στενά την ε, ρωσική δραστηριότητα εκεί. Και για να μην ξεχάσω βεβαίω και την Ουκρανία. Υπάρχει κάποια αναβάθμιση των δραστηριοτήτων ε, όσον αφορά την συνεργασία ε, στο στρατιωτικό τομέα με την ε, Ουκρανία. Thank you and uh, thank you for coming to the committee. Ευχαριστούμε Υπουργέ για την παρουσία σας. Για ορισμένα από αυτά από τα θέματα που αναφέρατε είναι βεβαίως η ΠΕΣΚΟ. Και μιλήσατε βεβαίως και για τα προγράμματα που υλοποιούνται. Ότι πολύ γρήγορα ολοκληρώσαμε την ΠΕΣΚΟ και, και, και καταρτήσαμε και τα προγράμματα. Έχετε κάποιες σκέψεις ωστόσο για την κατάρτιση πιο μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ε, υπό την ΠΕΣΚΟ που θα αποφασιστούν στο, στη, στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε ε, περισσότερες πληροφορίες ε, και σκέψεις για, τον, για τον λαϊκισμό και τις σχετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες στο τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα ε, να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς αυτό κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας. Ευχαριστώ κύριο Σπίτσουλα. Ευχαριστώ και εγώ να καλωσορίσω τον ε, Αντιστράτηγο και Υπουργό. Σας εύχομαι βεβαίως κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Και ε, ξέρω ότι και η δική μου χώρα θα βρεθεί στην ίδια θέση με εσάς, η Κροατία. Η Κροατία λοιπόν, η χώρα μου, ε, βρίσκεται στα Δυτικά Βαλκάνια και ξέρουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μία από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Όσον αφορά την ενίσχυση των συνδέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα, με τα έξι κράτη της Δυτικής, ε, ε, των, Δυτικών Βαλκανίων, έχουμε θέσει συγκεκριμένου και κοινού στόχου. Με απότερο σκοπό να προσχωρήσουν όλε αυτέ οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά ε, παρόλα αυτά εφικτό. Και στον τομέα της άμυνας δεν μπορώ παρά να ε, σας επισημάνω στο πνεύμα και των ερωτήσεων του κύριου Γκάλερ και να σας θέσω στο ερώτημα. Τι πιστεύετε για την ρωσική και τουρκική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί έχουμε ε, παρατηρήσει και παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια πόσο δηλητηριώδης είναι η ρωσική και τουρκική παρέμβαση στην, ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχετε κατά νου ε, να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες, όχι για να εξαλείψετε βεβαίως την ε, συμμετοχή και την εμπλοκή αυτών των δύο χωρών, αλλά για να προστατεύσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντά της και τη δική της παρέμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Φανσολίκα. Ευχαριστώ, Υπουργέ, ορίσατε. Όπως είπατε, η συνεργασία με τον βόρειο γείτονά σας, τη Ρουμανία, σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ένας ε, συνάδελφός μας, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια πρωτοφανής ενίσχυση ε, των ρωσικών στρατιωτικών ικανοτήτων στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει ήδη τεράστια ανισορροπία μεταξύ των ικανοτήτων της Ρωσίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αφετέρου. Αυτό οφείλεται και στη συνθήκη του Μαντρό του 1936 που απαγορεύει σε ξένες δυνάμεις, σε σκάφη δηλαδή, να εισέρχονται ε, στη Μαύρη Θάλασσα για περισσότερες από 21 μέρες, συνολικός αριθμός κάθε στιγμή μπορεί να είναι έως 7 κτλ. κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Επίσης, το ΝΑΤΟ πρότεινε στην Τουρκία να συνεισφέρει ε, με πλοία στρατιωτικά προκειμένου να εξορροπιστεί η κατάσταση. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο και πιο ενεργά με αυτό το θέμα και νομίζω ότι η πρόταση της Ρουμανίας θα έπρεπε να είχε τύχει υποστήριξη από τους ε, συμμάχους μας γιατί διαφορετικά ε, θα είμαστε απροετοίμαστοι απέναντι σε μια ενδεχόμενη ε, ρωσική επιθετικότητα. Βλέπετε ότι οι Ρώσοι συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις, πυράβλους Ισκερντέμ, επιράβλους s ε, S-400. Τώρα ε, η Τουρκία και η Ελλάδα ε, έχουν παραγγείλει αντίστοιχους πυράβλους. Πρέπει η Δύση να αναλάβει δράση. Αν θέλουμε πραγματικά και θέλετε κι εσείς να, να επιβεβαιώσετε ότι η Βουλγαρία ανήκει στη Δύση και προωθεί τις αξίες της. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια ερωτήματα. Κύριε Αντιστράτηγε, Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για τις ε, προτεραιότητες ε, όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν μια σειρά από χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των, ε, της ρωσικής επιρροής και παρέμβασης είναι ένα από τα μόνιμα θέματα αυτό που μας απασχολεί, ε, από αυτά που μας απασχολούν, η ρωσική προπαγάνδα ε, στην πολιτική και στην κοινωνία. Στην περίπτωση μάλιστα μίας χώρας, της Σερβίας, με την οποία υπάρχει μια σειρά από, από θέματα συνεργασίας, και έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να φέρουμε αυτή τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι ο υψηλός βαθμός ε, στρατιωτικής συνεργασίας με την ε, Ρωσία. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας, η επιθετικότητα που έχει επιδείξει η Ρωσία, ε, τις ενέργειες, αλλά και την επιθετική στάση που τήρησε κατά την προσέρτηση της Κρυμαίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα, ε, θέματα υπόψη, α, και να μην ε, ξεχνούμε βεβαίως και τις ε, κοινέ επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Λευκορωσίας, Ρωσίας και Σερβίας και μάλιστα πολύ κοντά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε για να φέρετε πιο κοντά την Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι σκοπεύετε να κάνετε για να πείσετε τη Σερβία να μειώσει τον ε, βαθμό στρατιωτικής συνεργασίας της με την ε, Ρωσία. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νόμιζα ότι το να, είμαι στην, ε, να κάθομαι ενώπιον της ε, Αμυντικής Επιτροπής της Βουλγαρίας είναι το πιο δύσκολο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω. Όμως το να βρίσκομαι σε εσά στη δική σας ε, Επιτροπή Άμυνας, Υποεπιτροπή Άμυνας, είναι εξίσου δύσκολο. Θα ξεκινήσω με τις απαντήσεις για το συντονισμό όλων των ε, διαφορετικών ε, στρατιωτήτων. Σχέδιο ανάπτυξης εκατοτήτων, ε, συντονισμός της άμυνας, πέσκο, βιομηχανικό σχέδιο, αμυντικό βιομηχανικό σχέδιο. Υπάρχει μία αλληλουχία αν θέλουμε να εφαρμόσουμε το στρατιωτικό σχεδιασμό, ξεκινάμε με την απειλή, τα σενάρια, τις ε, δυνατότητες. Και μια και ζούμε σε ένα ε, γοργά εναλλασσόμενο περιβάλλον ασφαλείας και άμυνας, το να έχουμε παράλληλες διαδικασίες με διαφορετικές πρωτοβουλίες και η αναζήτηση του συντονισμού ανάμεσα σε αυτές είναι νομίζω η σωστή πολιτική σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αμφιλεγόμενα θέματα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να αναπτύξουμε, στο να αναπτύξουμε και την ΠΕΣΚΟ χωρίς να υποτιμήσουμε την ΚΑΡΤ. Γιατί? Εμείς δεν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια από το μηδέν. όλα τα κρατημέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εμπειρία από τον αμυντικό σχεδιασμό. Κάθε έθνος γνωρίζει ποιες είναι οι δικές του ε, δυνατότητες, ικανότητες, ε, τα κενά του και έχουμε αρχικά, αρχικό σχεδιασμό και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στρατιωτικές δυνάμεις για να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά. Από τη βουλγαρική εμπειρία στην επιλογή των σωστών προγραμμάτων ε, για να ενταχθούμε στην πρωτοβουλία, ας πούμε, ΠΕΣΚΟ, ήταν... Μία από τις βασικές απαιτήσεις ήταν η Βουλγαρία ε, να ηγηθεί στις, ε, σε εθνικό επίπεδο ε, σε, αυτές τις, σε αυτό το πράγμα. Και παράλληλα να συμμετάσχουμε σε άλλες αποστολές του ΝΑΤΟ, συλλογικά. Δηλαδή, το να συμμετάσχουμε ούτω ώστε να δημιουργηθούν συλλογικέ δυνατότητες και capabilities ε, είναι το, ο σωστότερο τρόπος. Γιατί δεν μπορεί, δεν μπορεί κανένα κράτος του ΝΑΤΟ να δώσει όλα αυτά τα χρήματα για να αποκτήσει από μόνο του τις απαραίτητες ε, ικανότητες. Σας ευχαριστώ επίσης που υπερψηφίσατε τον ε, κανονισμό, το σχετικό κανονισμό, γιατί ο κανονισμό επιτρέπει στα ευρωπαϊκά κονδύλια να δοθούν για την ανάπτυξη αμυντικών βιομηχανικών προγραμμάτων και αυτό θα είναι και ένας μοχλός για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στο ΝΑΤΟ. Ε, η τεράστια πρόκληση της Τουρκίας είναι το επόμενο θέμα. Η Τουρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής, ε, γειτόνους Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και γείτονα της Βουλγαρίας. μοιραζόμαστε θαλάσσια σύνορα και χερσαία σύνορα με την Τουρκία κοινέ θάλασσε δηλαδή και χερσαία σύνορα. Γι' αυτό η Προεδρία της Βουλγαρία εστιάζει στι σχέσει Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι παίζει ζωτικό ρόλο η Τουρκία ελέγχοντα τους, μεταναστευτικέ τις Από το Ιράκ και τη Συρία έχουν εκατομμύρια μεταναστών που μπήκαν στο τουρκικό έδαφος. Ε, είναι δύσκολο γείτονα, όχι μόνο για μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι το να κρατήσουμε ανοιχτό το, τον ανοιχτό διάλογο σε όλα τα επίπεδα είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη χώρα αυτή. Για τη Βουλγαρία, ε, από πλευρά Βουλγαρίας να σας πω ότι εκτιμούμε τις τουρκικές ε, υποσχέσεις και είναι σημαντικό να τηρηθούν αυτές οι υποσχέσει, ούτω ώστε να ελεγχθούν τα σύνορα ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Τουρκία και να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση. Η Ουκρανία είναι τεράστια πρόκληση, από την άλλη. Άλλο θέμα. Ουκρανία. Η κρίση προκλήθηκε από την ρωσική εισβολή στην Κρυμαία. Ε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα τα εσωτερικά της Ουκρανίας. Είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα που έβαλαν οι Ρώσοι στην ε, Ουκρανία. Μετά την ε, προσάρτηση της Κρυμαίας, η κατάσταση στην Ουκρανία, και το είπε κάποιος Ρουμάνος βουλευτής, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, γιατί πραγματικά υπάρχει μια ε, οικοδόμηση στρατιωτικών δυνάμεων στην Κρυμαία και προσπαθεί να, η Ρωσία να αλλάξει το στρατιωτικό συσχετισμό στη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία πολιτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να την υποστηρίξει με όλα τα μέσα που διαθέτει και φυσικά το ΝΑΤΟ θα πρέπει να παίξει γι' αυτό το ρόλο του. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την Ουκρανία για να αναπτύξει αμυντικές ικανότητες και να μεταρρυθμίσει τις αναπλές δυνάμεις της. Η ΠΕΣΚΟ. Μακρόπνο πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μία επιτυχία η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Υπάρχουν από κάποιους, κάποιες αμφιβολίες για την επιτυχία της, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Τη δουλειά που έχει κάνει η Βουλγαρία. Τους υπολογισμούς και τις αξιολογήσεις που κάναμε για να μπούμε σε αυτά τα τρία προγράμματα που ανέφερα προηγουμένως, δείχνουν ότι, ότι η ΠΕΣΚΟ μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τις ευρωπαϊκές ε, αμυντικές ε, δυνατότητες. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις ε, αμυντικές δυνατότητες. Το να βασιστεί μονάχα στην νατοική συλλογική άμυνα πολιτικά είναι λάθος. Αν το κάνουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες και τις πολιτικές φιλοδοξίες πολιτικέ φιλοδοξίε και απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να παίξει αυτόνομο ρόλο. Η στρατιωτική ισχύ δυστυχώ μετράει ακόμα. Και ο στρατιωτικό ανταγωνισμό αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν κάποιε χώρε, δεν θα έλεγα ότι είναι ανταγωνίστριε, ε, θα έλεγα ότι είναι αντίπαλε. Όπω η Ρωσία, η Κίνα και πολλέ άλλε χώρε οι οποίες εξυγχρονίζουν το, το στρατό τους, ακόμα και τις στρατιωτικές τους ικανότητες, που στην περίπτωση του εύξηνου πόντου θα αλλάξει τα δεδομένα, θα αλλάξει τη στρατιωτική, τη στρατηγική συγγνώμη, ισορροπία. Αν χάσουμε την τεχνολογική υπεροχή, αν χάσουμε την υπεροχή στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, θα βρεθούμε σε δινή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα, είμαστε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό η Βουλγαρική Προεδρία αφιερώνει ιδιαίτερη πολιτική προσοχή στην ΚΠΑ, στην Κοινή Πολιτική Ασφαλής και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρόνος περνά. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεις. Πρέπει να οργανωθούμε περισσότερο και να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο σε αποτελεσματικές επενδύσεις για να οικοδομήσουμε ε, μοντέρνες ε, ε τελευταίας τεχνολογίας ε, στρατιωτικές ικανότητες, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστές, αν θέλουμε να συμμετέχουμε στην ε, στρατιωτική στρατηγική ισορροπία στην Ευρώπη. Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ενδιαφέρουν πολύ τη Ρωσία και την Τουρκία. Η Ρωσία προσπαθεί να επανακτήσει την επιρροή της, την οποία έχασε λόγω της κατάρρευσης ε, της Σοβιετικής Ένωσης, του απεριταρχικού καθεστώτος που υποστήριζε. Τώρα όμως βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση της ιστορίας της και προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις χώρες που αποτέλεσαν στο παρελθόν δορυφόρου της. Για μας, μία από τις προτεραιότητε βεβαίω είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται πραγματικά στην καρδιά της Ευρώπης. Το να έχουμε δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια υπό την επιρροή μιας άλλης δύναμης μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πρέπει να δείξουμε στις κυβερνήσεις, στους ε, θεσμούς αλλά και στους πολίτες αυτών των χωρών ποια είναι η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μας ενδιαφέρουν και μας νοιάζουν. Και ο καλύτερος τρόπος για να τους πείσει για τις ευρωπαϊκές αξίες είναι προφανώς το να δημιουργήσεις κοινά οικονομικά προγράμματα. Ξέρετε πόσο σημαντική βασική προτεραιότητα είναι για τη Βουλγαρική Προεδρία η δημιουργία υποδομών, ε, δρόμων μεταφοράς, δικτύων, προκειμένου να συνδέσουμε αυτές τις χώρες οδικά και ενεργειακά μέσω μιας κοινή εφοδιαστικής αλυσίδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρουν αυτές οι, οι, οι έξι χώρες όμως πρέπει και εκείνες να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις, τις αναγκές στο εσωτερικό τους προκειμένου να κινηθούν ε, και να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα αποτελέσει βεβαίως και κριτήριο για την προσχώρησή τους στην Ένωση στο μέλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, η Ρωσία, η Ρωσία και η Τουρκία θα δράξουν αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσουν τη δική τους επιρροή για τους δικούς τους εθνικούς σκοπούς. Βεβαίως, και ενάντια στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Μαύρη Θάλασσα. Είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, και ο Ρουμάνο Ευρωβουλευτή, πόσο σημαντική είναι η Μαύρη Θάλασσα. Η Βουλγαρία πραγματικά ανησυχεί πολύ για την, την ισορροπία έτσι όπω έχει διαμορφωθεί ε, από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι η σωστή απάντηση έχει δοθεί από το ΝΑΤΟ. Εμείς υποστηρίζουμε την ε, ενισχυμένη και προσαρμοσμένη ε, παρουσία. Έχουμε πλέον περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Μαύρη Θάλασσα. Η Βουλγαρία δεν υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ε, τριμερούς ε, ναυτικής δύναμης μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας και ε, Τουρκίας γιατί ακόμα και αν ε, δημιουργηθεί ένας τέτοιο στόλος δεν θα αλλάξει η ισορροπία. Χρειαζόμαστε το ε, το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, όχι τις ενέργειες μεμονωμένων ε, χωρών, ακόμη και αν συνεργάζονται. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Κοιτάξτε, τα στρατιωτικά πλοία των τριών χωρών αυτών που ανέφερα στο σύνολό τους είναι πολύ λιγότερα από τα ρωσικά πλοία. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ, την παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, που βεβαίως υπάρχει σε έναν βαθμό, αλλά χρειάζεται να συστηματικοποιηθεί και να, ενταθεί. Όσον αφορά τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Ρουμανία, ε, έχουμε προχωρήσει σε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία με επικεφαλή στη τη Ρουμανία, που περιλαμβάνει και ναυτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Και κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση ό,τι περνά από το χέρι μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Βουλγαρία ε, υποστηρίζει την ε, επιχειρησιακή μονάδα της Νοτιαλικής Ευρώπης και εμείς συμμετέχουμε με μια σειρά αποτάγματα, στρατεύματα ε, στην, στην, στις εξτρατήσεις και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Βεβαίως για το μέλλον αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Μαύρη Θάλασσα, που βεβαίω δεν έρχεται σε αντίθεση με την, ε, με την συνεργασία των τριών αυτών χωρών. Ρωσική προπαγάνδα. Νομίζω ότι η ρωσική προπαγάνδα βασίζεται πραγματικά ε, στις ψευδείς ειδήσει. Το κάνουν και στη χώρα μου. Προσπαθούν να επηρεάσουν τοπικές προεδρικές εκλογές στην ε, Βουλγαρία. Το έχουν κάνει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες αυτό. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει τα σωστά μέτρα καθώς έχει δημιουργήσει ένα σώμα εμπειρογνωμόνων που θα κληθούν ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες ε, δραστηριότητες προπαγάνδας και βεβαίω και σε αυτόν τον τομέα χρειαζόμαστε συντονισμένη απάντηση. Χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό. Όχι μόνο μέσα από δημόσιους φορείς, αλλά και με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών. Εταιρείε που ασχολούνται με την τεχνολογία προφορικής, που θα μπορέσουν να μας υποστηρίξουν και να μας συνδράμουν στο να εντοπίζουμε, να ανοιχνεύουμε τέτοιες ψευδείς ειδήσει που πραγματικά διαβρώνουν το ηθικό των Ευρωπαίων πολιτών και δημιουργούν μια αίσθηση έλλειψης ικανοποίησης, απεσιοδοξίας απέναντι στην πολιτική ηγεσία και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τη φιλοδοξία και την επιδίωξη της Ρωσίας να ε, ε, νικήσει και να ε, καταβαραθρώσει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες προκειμένου να ε, εγκαταστήσει απολυταρχικά καθεστώτα στην Ήπειρο. Ξέρετε ότι τέτοιου είδους σχέδια απολυταρχικά δεν στέφονται με επιτυχία μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί, αλλά ποτέ δεν δημιουργούν καλές σχέσεις με τους πολίτες τους. Και αυτό είναι που αυτό, αυτό είναι που, υπονομεύει τα καθεστώτα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να υπερασπιστεί τις αξίες της ε, στην καθημερινότητα των, ε, της ζωής των πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην ΑΠΑΤ μια άσκηση η οποία ε, ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Διαβάζοντας όμως το σενάριο, ε, είμαι βέβαιος ότι χρησιμοποιήθηκε ε, παραπλανητικά το σενάριο αυτό για να κρυφτούν οι πραγματικές προθέσεις που ήταν επιθετικές. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου θετικό στοιχείο καθώς ενισχύει την ένταση μεταξύ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Ρωσίας από την άλλη μεριά. Υπάρχει βεβαίως και ένας πολιτικός διάλογος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει όμως ο διάλογος αυτός να συνοδεύεται και από στρατηγική ικανότητα. Γι' αυτό και ο διάλογος, ε, αλλά και η, και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας είναι η καλύτερη απάντηση στι πολιτικέ που ακολουθεί η Ρωσία. Και τελευταίο ερώτημα για τη Σερβία. Η Σερβία πρέπει να αποφασίσει. Ναι, προσπαθεί να, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στι ευρωπαϊκές ε, αξίε, την ευρωπαϊκή προοπτική Αφενό και την, ε, τις φιλικές σχέσεις που παραδοσιακά έχει με τη Ρωσία. Εμάς μας ανησυχούν οι στρατιωτικές σχέσεις που έχει η Σερβία με τη Ρωσία. Είμαστε και γείτονε άλλωστε. Ε, μας ανησυχεί πάρα πολύ η προμηθεια μιτ MIT-29 από την ε, Σερβία. Από τη, ε, αγόρασε η Σερβία δηλαδή τα, τα συστήματα αυτά από τη Ρωσία. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε από το να πούμε, από το να πούμε στην ε, Σερβία ότι αν θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στι ευρωπαϊκέ στρατηγικέ επιχειρήσει και όχι στι ρωσικέ. Αυτό βεβαίω είναι εσωτερικό ζήτημα τη Σερβία. Εμεί απολύτω βεβαίω θα συνεχίσουμε τον διάλογο με τη χώρα αυτή. Εμεί ω χώρα, ω Βουλγαρία, έχουμε και πολύ καλέ στρατιωτικέ ε, σχέσει με την Σερβία πολύ συχνά συμμετέχουν σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις ε, σε ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος της Βουλγαρίας και είναι πάντοτε αυτές οι επιχειρήσεις μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να έρχονται σε επαφή οι ένοπλες δυνάμεις του, χωρών του ΝΑΤΟ με τις ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας προκειμένου να έρχονται και να, και δημιουργείται και μια... να δημιουργούνται και πρακτικές εμπειρίες ε, στους αξιωματικούς του Σερβικού στρατού και όλα αυτά πάντοτε λειτουργούν και ως μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθήσει κανείς ε, και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για να τονώσει, να τονίσει μάλλον το, την ευρωπαϊκή προοπτική της ε, Σερβίας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Όχι, λέει η πρόεδρο, δεν υπήρχαν άλλε παρατηρήσει. Αν με επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ήθελα να κάνω και κάποιε άλλε ερωτήσει ε, που σχετίζονται επίση με τα Δυτικά Βαλκάνια και εν μέρη με την ευρύτερη γειτονία του. στις διαβουλεύσεις μας με τους ε, εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υψηλού επίπεδου. Μάθαμε για τα πιλωτικά έργα που τρέχουν σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, μεταξύ ΝΑΤΟ δηλαδή και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Χώρες όπως ε, η Βοσνία Ζεγοβίνη, η Μολδαβία, η Τινησία αναφέρθηκαν ως ε, πιλωτικές περιοχές για τέτοιου είδους συνεργασία. Θέλετε να μας πείτε κάποιες σκέψεις ε, για αυτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Το επόμενο θέμα είναι η στρατιωτική κινητικότητα και φυσικά και εδώ υπάρχει περιθώριο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. μετά από τη διακήρυξη της Βαρσοβίας ε, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εξελίξεις στον τομέα αυτών. Uh, thank you, ma'am. Uh, cyber security project. Uh, cyber security is uh, Λοιπόν, για αυτά που αναφέρατε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, το ΝΑΤΟ ουσιαστικά αποφάσισε ότι ο τομέας του κυβερνοχώρου είναι ο πέμπτος ε, τομέας ε, ε, στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Δραστηριοτήτων μάχης, δηλαδή. Ο κυβερνοχώρος, δηλαδή, θα αποτελέσει στο μέλλον χώρο πολέμου. αλλά είναι και χώρος ε, σημερινών πολέμων. Διότι καθημερινά παρατηρούμε δραστηριότητες ε, τέτοιου είδους ε, στον κυβερνοχώρο. Αναφέρομαι σε δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο σχεδιασμένες για να περιλαμβάνουν και χώρες εταίρους. Διότι υπάρχουν δύο οδοί στο ΝΑΤΟ, η εσωτερική οδός της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και του σχεδιασμού στον κυβερνοχώρο και λόγω αυτού του κυβερνοχώρου ως χώρου πολέμου, ως χώρου μάχης, ως πεδίου μάχης, το ΝΑΤΟ ουσιαστικά αποφάσισε να υλοποιήσει το σχεδιασμό στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, του, σχεδιασμού, του αμυντικού σχεδιασμού, οικοδόμηση δηλαδή δυνατοτήτων αμυντικών, ε, αλλά και να ενσωματώσει το σχεδιασμό στον κυβερνοχώρο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της άσκησης υλοποιεί το ΝΑΤΟ μέτρα άμυνα στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο αυτής της άσκησης. Αυτή είναι η εσωτερική οδός. Η εξωτερική οδός φυσικά είναι η συνεργασία με χώρες εταίρους. Διότι για να επιτύχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του κυβερνοχώρου χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερες φιλικές χώρες στο πλευρό μας. Χρειάζεται να υλοποιήσουμε κοινά μέτρα προστασίας ημών, αλλά και για να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πρόκειται, πιστεύω, για μια θεμητή πολιτική απόφαση το να συμμετέχουν και εταίροι στη μάχη αυτή κατά των ε, δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του πολέμου θα έλεγα μάλιστα στον κυβερνοχώρο που μένετε ακόμη ήδη σήμερα. Η στρατιωτική κινητικότητα, ναι, πράγματι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική η στρατιωτική κινητικότητα, όχι για την άμυνα τη Ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά και για τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική, στρατιωτική κινητικότητα πιστεύω αποτελεί το τέλειο παράδειγμα του πώ ε, μπορούν να συνεργαστούν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντα υπόψη ότι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει τη κινητικότητα ε, είναι ε, η εσωτερική συνεργασία στις ε, χώρες ε, που αποτελεί αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων, ζήτημα που μπορεί να επιληθεί μόνο από κοινή συνεργασία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και όχι μόνο από τον ένα ή από τον άλλο. Πιστεύουμε ότι εμείς ως Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να αισθανόμαστε αισιοδοξία για το project αυτό ε, και 28 χώρες ε, ε, συμμετέχουν σε αυτό το project και έτσι σε όλους τους τομείς του ζητήματος αυτού, της ε, στρατιωτικής κινητικότητας, της διέλευσης των συνόρων, βλέπουμε να εμπλέκεται η συνοριοφυλακή, τα συστήματα μεταφοράς, κάποιες φορολογικές αρχές, που ελέγχουν την κυκλοφορία αγαθών και προσώπων ε, διασυνοριακά. Το project αυτό ουσιαστικά θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμβολή στην κοινή ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Διότι θα μας επιτρέψει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα, να μετακινούμε με μεγάλη ταχύτητα ε, υλικό στρατιωτικό από τη μια χώρα στην άλλη, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ε, όπου συνεπάγεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους, αλλά και για την περίπτωση στρατιωτικής εκπαίδευσης. Μπορούμε να μετακινήσουμε στρατεύματα για σκοπούς αποτροπής, αποθάρρυνσης πιθανών αντιπάλων μας από επίθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλέ οι τελευταίες παρατηρήσεις ω εισαγωγή στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξη, που είναι ένα που έχει πέντε ομιλητές για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για την επιχειρησιακή κινητικότητα με πέντε ομιλητέ, όπω είπα, το πάνελ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Άμυνα της Βουλγαρίας ε, που συμμετείχε στις ε, συζητήσεις μας. Ο Υφυπουργό συνοδεύτηκε από μια ολόκληρη αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ όλους για τις απόψει σα για αυτή την εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και καλή τύχη για την Προεδρία σας. Ελπίζω να είναι επιτυχής βασίζεστε, Μπορείτε να βασιστείτε στην ε, βοήθειά μας και σας παρακαλώ ας χειροκροτήσουμε όλοι τον Υφυπουργό. Thank you. Παραμείνετε στην αίθουσα παρακαλώ, θα περάσουμε πάρα αυτά στο επόμενο σημείο. Καλώς ορίσατε στην συζήτηση αυτή που θα κάνουμε. Ε, είναι το τελευταίο σημείο της ε, πρωινής συνεδρίασης. Είναι ένα θέμα για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για την στρατιωτική κινητικότητα. Έχουμε πολλοί αριθμούς πανελίστες Να σας παρουσιάσω τους εκπροσώπους δύο σημαντικών Ινστιτούτων, τον κύριο Αγνό, ε, τον κύριο Αγνό Μολινάρ, εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο οποίος θα μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εν συνεχεία, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Τη Reuters της Γενικής Διεύθυνσης MOVE. Μετά έχουμε ανώτατους εκπροσώπους ε, του ΝΑΤΟ, ανώτατους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, τον Τίμο Κόστνερ, ε, διευθυντής, τον ξέρετε, Έχει ξανάρθει στην Επιτροπή μας, έχει μιλήσει εκπροσωπώντας τον ΝΑΤΟ Επίσης, έχουμε έναν ανώτατο αξιωματούχο και υπεύθυνο όλης αυτής της προσπάθειας, το κύριος Hans van Santen, υποδιευθυντής διεθνών υποθέσεων του Υπουργείου Άμυνας της Ολλανδίας. Και το τελευταίο, αλλά σημαντικότατο εκπρόσωπο, εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Αμυντικής, ε, του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού, τον κύριο Ζων Γιούρι Μαχτή. Και αυτός έχει ξανάρθει στην Επιτροπή μας. Έχει επισκεφθεί πολλές φορές την υποεπιτροπή μας, Εκπροσωπώντα την EDA. και εκπροσωπώντα τον ε, εκτελεστικό διευθυντή του, της EDA, του Ευρωπαϊκού Ομιλικού Οργανισμού. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, συνάδελφοι, και χωρίς ε, χρόνο τριβή. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Αγνό Μολινάρ για να παρουσιάσει τη δική του σκοπιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια εισαγωγικά λόγια θέλω να πω για το θέμα της κινητικότητας, της στρατιωτικής κινητικότητας, γιατί είναι επίκαιρο και συνεχεία να περάσω στη διαδικασία και να δώσω το λόγο ε, στους υπόλοιπους συναδέλφους του πάνελ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει τις, και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στις ανάγκε του. Εντάσσεται στο ευρύτερο θεματολόγιο τη Ένωση, στα πλαίσια τη Παγκόσμια Στρατηγική, για να ενισχύσει την ασφάλεια και άμυνα και να προστατεύσει τα συμφέροντα τη Ένωση σε ένα πολύ πιο προβληματικό ε, περιβάλλον ασφάλεια. Θέλει να διευκολύνει και να ε, επιταχύνει την εξωτερική ανάπτυξη και εσωτερική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ε, υλικού και ανθρώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη, μπήκε πέρυσι, όταν κάποια κράτη-μέλη χτύπησαν τον κόδωνα κινδύνου μετά τις εμπειρίες που είχαν για τα φυσικά και κανονιστικά φράγματα που εμποδίζουν την διασυνοριακή μετακίνηση και επομένως μειώνουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει από κοινού και αυξάνει το κόστος βεβαίως και τα σημεία που είναι ευάλωτα, πρωτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φυσικά είναι περίπλοκος ο τομέας, για να δουλέψουμε και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην παρουσία πολλών ομιλητών εδώ με ειδικέ αρμοδιότητε και καταρχά πρέπει να σεβαστούμε την εθνική κυριαρχία για τη μετακίνηση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων που θα περνούν από την ε, εθνική μα επικράτεια. Δεύτερον, ε, είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Ε, έχει να κάνει όχι με τα αμυντικά θέματα, μεταφορών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει, είναι πολύ διάστατο. Μιλάμε για μετακινήσεις ε, από αέρος, θάλασσας και ξηρά ε, με τους ειδικού τρόπους μεταφοράς, με τα ειδικά θέματα και τους ε, ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενου κάθε φορά. Κάτι άλλο που περιπλέκει τα πράγματα. Φυσικά θέλει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο στόχο τη. Παράλληλα, θα πρέπει να κάνει στενό διάλογο με του εταίρου ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του σημαντικού εταίρου, ε, στα πλαίσια αμοιβαία ενίσχυση και συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ κάνει πολλή προσπάθεια στον τομέα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικά εργαλεία όμω στη διαθεσή τη που δεν έχει το ΝΑΤΟ και τελικά ε, η πιο αποτελεσματική λύση μπορεί να βρεθεί μόνο ε, με τη συνεργασία. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές ε, που διέπουν ε, αυτή την επιχείρηση. Υπάρχει και ε, ένα κλασικό πολιτικό και αμυντικό και πρακτικό θέμα. οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τα λοιπά και θα μπορεί να είναι και διμερός και μέσω του ΝΑΤΟ. Οι συνάδελφοι θα συμπληρώσουν αυτά που λέω εγώ αλλά μέσα από το πλαίσιο EDA ε, ε, έχει εγκύψει ε, πολλών θεμάτων πολλά, επί πολλά χρόνια. Μετά από αιτήματα πολλών κρατών μελών έχει δημιουργήσει και ομάδες ad hoc και φανταζόμαι ότι ο εκπρόσωπος της EDA θα σας ενημερώσει για αυτό, το πράγμα. 10 ε, Οκτωβρίου του 2007 υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση της Μογκερίνη και της Κομισιόν για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το πλαίσιο για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Τρεις βασικοί τομείς ε, εργασίας εντοπίστηκαν. Ε, θέματα υποδομών, το θέμα που αφορά τους ε, κανόνες, κανονισμούς, ε, νομικά θέματα, καθώς και οι κυβερνοαπειλές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε να προωθήσουμε με βάση τις στρατιωτικές ανάγκες που θα καθορίσουν τα κράτη-μέλη. Το επόμενο βήμα είναι η, η Κομισιόν και είπατε Εκπρόσωπος να ετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης μέχρι τον Μάρτιο του 2018 που θα βασίζεται στα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων ad hoc στα πλαίσια, που εργάζονται στα πλαίσια της CDA. Το Δεκέμβριο του 2017 τα κράτη-μέλη συμμετείχαν στην ΠΕΣΚΟ, Νοέμβριο και Δεκέμβριο μάλιστα. Όσα κράτη-μέλη συμμετείχαν στην ΠΕΣΚΟ εντόπισαν την ανάγκη για να προωθηθούν κάποια project, ούτω ώστε να υπάρχουν κάποιες ε, σαφέστερες δεσμεύσει. Ε, σε αυτό το πλαίσιο. Η Ολλανδία είναι η πρώτη χώρα που θα ηγηθεί και ο Hans Van Santen θα σας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποφάσισαν το Δεκέμβριο του 2017 ε, μέσω μιας κοινή δήλωση να υπάρχει ε, να δοθεί προτεραιότητα στη στρατιωτική κινητικότητα. Κατά την άποψή μου, ε, η βασική δουλειά τώρα είναι η δουλειά που κάνουν τα, οι ομάδε ad hoc τη EDA και θα είναι η βάση ε, του σχεδίου δράση που θα παρουσιάσει η Κομισιόν και η Πατή Εκπρόσωπο. Αυτή η δουλειά γίνεται με τρόπο που δεν έχει αποκλεισμού, με χαρτογράφηση των προβλημάτων. Ε, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι να υποστηρίξει την ύπατη εκπρόσωπο σε όλε αυτέ τι προσπάθειε και να συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο σε μια συνεκτική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς και τα θεσμικά όργανα ε, και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για να προωθήσουμε ε, μια συντονισμένη απάντηση follow-up ε, με, στα πλαίσια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες μας που έχουμε στον τομέα. Τέλος, τελευταίο σχόλιο. Φυσικά η υπηρεσία μου, η υπηρεσία εξωτερική δράση, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Υποεπιτροπή σα ε, για να προχωρήσουμε, καθώς θα ασχολούμαστε περαιτέρω με το θέμα ε, και περιμένω τις ερωτήσεις σας, στις οποίες θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μολινάρ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, διευθυντή κύριο Reuters της Γενικής Διεύθυνσης MOVE, αν και γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι ε, ενωσιακή αρμοδιότητα, ούτε θέλουμε να υπονομεύσουμε την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε αυτό το, σε αυτό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Η ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης είναι προτεραιότητα και στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί έως το 2025 μια πλήρης ένα πλήρες ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας ε, προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό ταχαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κάτι τέτοιο απαιτεί την άρση πρακτικών νομικών εμποδίων και τα ζητήματα της στρατηγικής κινητικότητας ε, άπτονται και του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπάρχουν λοιπόν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία δυνατότητες να ενισχυθεί η στρατηγική κινητικότητα. Όπως είπε ο κύριος Μολινάρ, τον Οκτώβριο η Κομισιόν και η ύπατη εκπρόσωπος ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για τους βασικούς τομείς ε, στους οποίους θα μπορούσαν να αναλυθούν δράσεις για να ενισχυθεί η στρατιωτική κινητικότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η χρήση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, η ενίσχυση των ε, επενδύσεων, ρυθμιστικά και κανονιστικά ζητήματα όπως είναι τα τελωνιακά θέματα καθώς και η συνεργασία στην αντιμετώπιση βρυθικών απελών ορίζει και ορισμένους στόχους και ορισμένα βήματα για το, για το επόμενο διάστημα. Βάσει του έργου που έχουν επιτελέσει τα κράτη-μέλη και θα, με χαρά θα ακούσω και τον κύριο Βαν Σάντεν μετά, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, της συνεργασίας ε, της ΕΕΔ και του ΝΑΤΟ, η ύπατη εκπρόσωπος και η Κομισιόν θα υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική κινητικότητα το Μάρτιο του 2018. Και αυτό όπως τονίσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ε, θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη. Εκεί θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένε δράσεις με συγκεκριμένους, από συγκεκριμένου φορείς, οι οποίοι συμπληρωματικά θα συνεργάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα των ε, υποδομών μεταφορών, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης MOVE, το βασικό καθήκον είναι να προσδιοριστούν οι απαιτήσει που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας και βέβαια αυτό ε, κατά κύριο λόγο θα γίνει από την ίδια τη στρατιωτική κινητικότητα. Σε δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να ε, συγκρίνουμε τις στρατιωτικές ε, απαιτήσει με τις παραμέτρους 10T, να εντοπίσουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένες και να διαπιστώσουμε αν τα TEN-T που έχουν ήδη ε, καθιερωθεί ε, είναι κατάλληλα και για στρατιωτικούς σκοπούς και αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά. Και έπειτα, μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, τον προσδιορισμό των ελλείψεων και τη χαρτογράφηση που θα κάνουμε, θα χρειαστεί να προχωρήσουμε και στον προσδιορισμό των αναγκαίων επενδύσεων για στρατηγικούς σκοπούς που ε, απαιτούνται. Και να τονίσω βεβαίω ότι γι αυτό, ε, μπορεί να, αυτό μπορεί να χρησιμεύσει και για μη στρατιωτικού σκοπούς. Και το τελευταίο βήμα είναι να ποσοτικοποιήσουμε βεβαίω και το κόστο. Κατά αυτή την έννοια, αυτή η ιδέουσα χρήση των υποδομών θα ωφελήσει όλα τα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα θα ενισχύσει και θα διευκολύνει και τη στρατιωτική κινητικότητα. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες μετά την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου δράσης ε, ώστε να έρθω και να σας ενημερώσω σχετικά με τις δράσεις αυτές, τις πρωτοβουλίες, αλλά και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με όλους τους φορείς στον τομέα, ε, που σε μεγάλο βαθμό μάλιστα δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Θα έχουμε... Ε, Όμω η αξιοποίηση τη ήδη ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια κατεύθυνση και στην δημιουργία, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας πραγματικής αμυντικής ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίσε και ο πρόεδρο Γιούγκερ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Το θέμα είναι καυτό. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε την επιθετικότητα της Ρωσίας ε, απέναντι στην Ουκρατία, ε, στην Ουκρανία, την προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά και την ανάπτυξη του Ανατολικού Βραχίωνα του ΝΑΤΟ. Ανέκυψαν πραγματικά, πρακτικά προβλήματα ε, όσον αφορά την ανάπτυξη νατοικών δυνάμεων στις βαλτικές χώρες και έχουμε συγκεκριμένες ε, θέσεις και σκέψεις, προβληματισμούς ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, την ειδική προσοχή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Είναι πολύ ευρύτερο λοιπόν το, το, το θέμα ε, από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια ε, και με πολύ μεγαλύτερη θέρμη συζητείται πλέον εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε άλλωστε διαπιστώσει και με την ευκαιρία επισκέψεων που έχει πραγματοποιήσει η υποεπιτροπή μας ε, ε τους ε, τις διάφορες μορφές που λαμβάνει η στρατιωτική συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ε, σε όλες αυτές τις περιοχές τις οποίες έχουμε επισκεφτεί. Διευθυντά, κύριε Κώστερ, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ μαζί μας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις ε, με την Επιτροπή σας. Η Πρόεδρος ε, παρουσίασε ήδη το υπόβαθρο, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της ασφάλειας που σίγουρα αποτελεί την για τη δική μας ε, μεταβολή ε, της στρατιωτικής κατάστασης και ως αποτέλεσμα την εξέταση του ζητήματος της στρατιωτικής κινητικότητας. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο οι ρωσικές δραστηριότητες ανατολικά. Όταν αναφερόμαστε στη στρατιωτική κινητικότητα στο ΝΑΤΟ, αναφερόμαστε εξίσου και στη μετακίνηση προς άλλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα προς τον Νότο, όπου έχουμε μια τεράστια ζώνη αστάθειας και ανασφάλειας. Επίσης αφορά και τη δυνατότητα μετακίνησης στρατευμάτων και εξοπλισμού και πέραν του Ατλαντικού, διότι εκεί έχουμε και συμμάχου. Ε, τον ένα σύμμαχο που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχο στρατευμάτων μάλιστα. Η στρατιωτική κινητικότητα λοιπόν ορίζεται από εμάς ως μια βασική απέτηση ταχείας ε, ε, κινητοποίηση σε μια σύνοδο κορυφής του 2016 στη Βαρσοβία οι ηγέτες μας ανέφεραν τη στρατιωτική κατάσταση παρουσία του ΝΑΤΟ με μια ε, μέτρια παρουσία στην Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες της Βαλτικής, στην Πολωνία, μια περιορισμένη παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα. Μια μέτρια λοιπόν παρουσία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ταχείας ε, κινητοποίησης ε, της περιορισμένης αυτής παρουσίας. Μιλάμε τώρα όχι μόνο για τις μαγωγικές μονάδες, αλλά και για τις αμυντικές μονάδες των χωρών, των εν χωρών. Ενισχυμένες με τις μάχημες ομάδες που υπάρχουν εκεί και μερικές φορές και με την παρουσία των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ε, EDI, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής, ε, ε, που ονομαζόταν ERI, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία διαβεβαίωσης, διασφάλισης, αλλά όλα αυτά έχουν αξιοπιστία ως αποτρεπτικό μέσα, μόνο αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις, ε, τα στρατεύματά μας και κυρίως τον βαρύ εξοπλισμό γρήγορα και εντό ε, των χρονικών περιθωρίων που έχουμε ορίσει στα σχέδια που έχουμε προετοιμάσει εκ των προτέρων. Ο εξοπλισμός μετακινείται πιο δύσκολα από ότι ε, τα στρατεύματα, η ΖΙΤΖΕΤ και η ΡΑΝΕΡΑ και μετακινούν πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη καθημερινά, οπότε η μεταφορά ανθρώπων και προσωπικού δηλαδή δεν είναι ότι πιο δύσκολο. Δεν είναι το πιο δύσκολο. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι κινήσει που προβλέπουμε κατά κύριο λόγο θα πρέπει να γίνονται σε εποχέ ειρήνη. Τα μέτρα λοιπόν που λαμβάνουμε και η πρόσβαση στην οποία χρειαζόμαστε πρόσβαση και η νομοθεσία που υλοποιούμε ε, βασίζονται στην ε, αντίληψη ότι όλα γίνονται σε εποχή ειρήνης, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νομοθεσία που θα έχουμε για εποχές κρίσης, ε, δεν μπορούμε να στρατολογήσουμε εξοπλισμό μόνο για εποχές κρίσης. Οπότε σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι ό,τι έχουμε υποδειχθεί ότι λειτουργεί σε εποχές ειρήνης. Και έχουμε εντοπίσει τον ΝΑΤΟ τέσσερις τομείς ε, που χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Ε, οι άλλοι ομιλητές ε, ήδη αναφέρθηκαν σε αυτούς. Χρειαζόμαστε δουλειά σε θέματα υποδομής, νομοθεσίας και διαδικασιών διασυνοριακά και για τη διέλευση των συνόρων. Επίσης χρειάζεται να αυξήσουμε τις δυνατότητες μεταφοράς, αερομεταφοράς και πρέπει να προσαρμόζουμε το διοίκησή μας και τον έλεγχό μας για τη διοικητική μέρημνα. Ε, σε θέματα υποδομής, ε, το είπε ήδη ο συνάδελφος, ε, η υποδομή πρέπει σε όλη την Ευρώπη και εδώ δεν μιλάμε μόνο για δρόμους, μιλάμε για δρόμους, υδροδρόμους, υδατινές οδούς κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα χειρισμού των ροών στρατιωτικού εξοπλισμού και βαρέως εξοπλισμού. Είναι σημαντικό οι γέφυρες να είναι αρκετά ε, ανθεκτικές, να είναι αρκετά πλατιές οι κτλ. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τις προδιαγραφέ που έχουμε στον ΝΑΤΟ, είναι και ο τρόπος που σχεδιάζει κανεί που κατασκευάζει συγκεκριμένε υποδομέ. ώστε η ροή των δυνάμεων και του εξοπλισμού να είναι απρόσκοπτη. Επίσης έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε επίγνωση της κατάστασης δεν αφορά άμεσες εργασίες σε γέφυρε και σε δρόμους. Ξεκινάμε τη χαρτογράφηση της, ε, των υποδομών. Και στο ΝΑΤΟ γνωρίζουμε ελάχιστα ουσιαστικά για οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του Βερολίνου. Γιατί? διότι το παλιό καιρό ήταν κομμάτι του Σύμφωνου της Βαρσοβίας και μετά από το 1990 τα άλλαξε η κατάσταση σαφώ. δεν αισθανθήκαμε ε, άμεση ανάγκη χαρτογράφησης των υποδομών και να υλοποιήσουμε τα ίδια. Είχαμε τα, τα ίδια σχέδια που είχαμε και κατά τον ψυχρό πόλεμο. Και θα θυμάστε ότι για τουλάχιστον δύο δεκαετίε η Ρωσία ανέπτυσε, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε εμεί, ε, αναπτύχθηκε, αναπτυσσόταν ω ε, στρατηγικό εταίρο του ΝΑΤΟ αντί για σαφή ανταγωνιστή. Οπότε τι προσπαθούμε να κάνουμε, να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η κατάσταση της υποδομής, των υποδομών στην Ανατολική Ευρώπη. Δεύτερον, να την αναβαθμίσουμε και ο κ. Μισράτος το είπε πολύ σαφώς ε, τι είναι κοινό συμφέρον ε, και ενδεχομένω κοινή προσπάθεια μεταξύ ε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μορφή θα μπορούσε να έχει, έχουμε τα στρατιωτικέ προδιαγραφέ και απαιτήσει στα σχετικά στάνταρ, εφόσον ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα επιμέρου κράτη-μέλη, του συμμάχου, αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα την κατάσταση ω περαιτέρω βήμα, διότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κατασκευαστική εταιρεία όπω γνωρίζετε. Χρησιμοποιούμε μόνο ε, μη στρατιωτικέ υποδομέ ε, και μόνο όταν χρειάζεται. Όσον αφορά τι νομοθετικέ διαδικασίε, ε, και πάλι εδώ υπάρχει ένα κοινό συμφέρον ε, να γίνει μια κοινή προσπάθεια με το EDA. έχουμε κάποιε διαδικασίε ήδη. Έχουμε ήδη καταφέρει να πείσουμε τους επιμέρους συμμάχους να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία ώστε να υπάρχουν ε, διπλωματικές άδειε για συγκεκριμένα επικίνδυνα προϊόντα, για πυρομαχικά, πιο γρήγορα, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για νομοθεσία εθνικού επίπεδου, μιλάμε και για διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ε, κυριολεκτικά μέχρι και τα σύνορα ε, και πρέπει να έχουμε απλά πράγματα όπως έντυπα ηλεκτρονικά τα οποία να λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα, να διεκπεραιώνονται γρήγορα και απρόσκοπτα εύκολα. Ε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και βρισκόμαστε σε συνομιλίε με την NDA για να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη λύση, ποιο θα κάνει τι. Και πιστεύω ότι έτσι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πολύ γρήγορα πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Ε, τρίτη κατηγορία, οι δυνατότητε οι μεταφορικές. Δεν έχουμε αρκετά αεροπλάνα, τρένα και οχήματα για να μεταφέρουμε προσωπικό και εξοπλισμό γρήγορα. Οπότε απαιτούνται πολλές ε, επενδύσεις. Στο ΝΑΤΟ έχουμε τη διαδικασία σχεδιασμού, αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ που έχει συγκεκριμένους στόχους δυναμικού ε, για τους συμμάχους και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι έχουν τους ε, στόχους δυναμικού, τους γνωρίζουν και ότι τους υλοποιούν γρήγορα, ώστε να έχουν μεγαλύτερες μεταφορικές δυνατότητες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση ε, στον ιδιωτικό τομέα, διότι πολλές κινήσεις διευκολύνονται σήμερα από ε, ιδιωτικούς, από διώτες αναδόχους, κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό. Ε, για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στο Αφγανιστάν σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετήθηκε από αναδόχους ιδιώτες. Αλλά οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ε, πρόσβαση σε πλοία ρορό, σε τρένα κτλ. Ε, και μετά πρέπει, εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες γιατί οι υποδομές, ε, το τροχείο υλικό σήμερα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, δεν είναι κομμάτι κρατική ιδιοκτησία, πολλέ φορέ είναι ιδιωτική ιδιοκτησία. Και δεν μπορούμε να ξεκινάμε να συνάπτουμε τι συμβάσει μόλι εμφανιστεί η κρίση. Πρέπει να υπάρχουν συμβάσει από πριν. Πολύ καιρό πριν, οπότε απαιτούνται κάποιε προσπάθειε. Τέλο, ε, διοίκηση και έλεγχο. Η διοικητική μέρημνα ίσω είναι ένας από τους τομεί ε, όπου χρειάστηκε να περικόψουμε περισσότερο τις στρατιωτικέ μας δομές ε, κατά την δεκαετία των αμυντικών περικοπών. Σήμερα προσαρμόζουμε την στρατιωτική δομή που έχουμε στο ΝΑΤΟ και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της δομής είναι το να επαναφέρουμε σε μεγάλο βαθμό την διοίκηση και τον έλεγχο της διοικητικής μέρημνας. Και ειδικότερα στο επίπεδο του κοινού επιτελείου έχουμε μονάδες διοικητικής ε, μέρημνας, τις ονομάζουμε επιτελείο διοικητικής μέρημνας, που διευκολύνουν, οργανών και συντονίζουν την κίνηση, τη ροή των δυνάμεων εντός και ε, κατά μήκο της Ευρώπης. Και ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά αυτής της δομής είναι ότι δημιουργούμε μία ολόκληρη ε, διοίκηση ε, των μετόπισθεν. Αυτά κάνουμε. Σε θέματα διοίκησης και ελέγχου έχουμε ήδη το σχεδιασμό και τη δομή. Η δομή αυτή ε, προβλέπουμε ότι θα επικυρωθεί από τους Υπουργούς Άμυνας το Φεβρουάριο και ελπίζουμε να κάνουμε τις τελικές ανακοινώσεις επί των λεπτομεριών για το ποια ε, επιτελεία θα πάνε πού μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου. Θα κλείσω εδώ, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό, το ανέφερε και ο κ. Μολενάρ. Ό,τι είπαμε αφορά πολλές κρατικές προσπάθειες. Ε, στο ΝΑΤΟ φυσικά συνεδριάζουν συνήθως Υπουργοί Άμυνα και συζητούν για την ε, στρατιωτική κινητικότητα κτλ. Αλλά η διέλευση συνόρων, ο συντονισμός των κινήσεων, η νομοθεσία, όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν ε, ελέγχονται μόνο από τους Υπουργού Άμυνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟ όσο και σε εθνικό επίπεδο να συνομιλούν άπαντες μεταξύ τους και για παράδειγμα οι Υπουργοί Μεταφορών κάθε χώρας να αντιλαμβάνονται τι απαιτήσει έχουν οι συναδελφοί του Υπουργοί Άμυνα ε, και τι επιθυμούν να γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσω εδώ. Είμαι ανοιχτό για ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τον Διευθυντή. Κυρίες και κύριοι, η Ολλανδία είναι σημαντική χώρα. Διαμορφώνει την έννοια της στρατιωτικής ε, κινητικότητας και μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον Hans Van Santen, αναπληρωτή Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων στο Τμήμα Πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας των Κάτω Χωρών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι είμαστε επικεφαλής σε ορισμένες προσπάθειες. Να σας εξηγήσω γιατί ξεκινήσαμε αυτό το project. Όλα ξεκινήσαν το 2017 όταν ο προηγούμενο ε, υπουργό Χάνες έγραψε μία επιστολή στην ύπατη εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη και στον εκτελεστικό διευθυντή της, ε, του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού, τον κύριο Ντομέκ, ε, λέγοντας ότι η ιδέα της στρατητική κινητικότητα ε, είναι ότι από την εμπειρία μας προκύπτει σε διάφορες ασκήσεις και σε διάφορες μετακινήσεις στην Ευρώπη ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και προσκόμματα, διάφορα κολλήματα, ε, τελωνία, υποδομές κλπ. Και μερικές φορές οδήγησε σε ορισμένε αυτοκινοπομπές να περιμένουν στα σύνορα επί εβδομάδες γιατί δεν μπορούσαν να διέλθουν τα σύνορα. Αυτό το θέμα το άκουσαν οι άλλοι, το άκουσε η κυρία Μογκερίνη, ε, ασχολήθηκε πολύ γρήγορα με το πρόβλημα αυτό και ασχοληθήκαμε με τρεις άξονες. Ο ένας είναι αυτός που έχει ξαναφερθεί, η ομάδα ad hoc ε, του Ευρωπαϊκού Μυντικού Οργανισμού. Χθες ολοκληρώσαμε μία έκθεση στα προβλήματα ε, που υπάρχουν στους διάφορους τομείς και αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη δράση για την ε, έκθεση δράσης που θα ετοιμάσει η Κομισιόν. Αυτό είναι ένας άξονας, ο οποίος πάει πολύ καλά τώρα. Ο δεύτερος είναι το project PESCO που έχει ήδη αναφερθεί. Ε, η στρατιωτική κινητικότητα στα πλαίσια της μόνιμης διαφορεμένης συνεργασίας είναι ένα από τα project. Ε, το πιο δημοφιλές. Έχουμε 24 συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Η αρχική συνεδρίαση θα γίνει 1η Μαρτίου και εκεί θα εστιάσουμε σε διάφορα θέματα που είναι κρεμή. Ε, πρέπει να δούμε την ατζέντα καταρχήν. Ε, η ιδέα είναι να συνεχίσουμε την πολιτική πίεση αυτή που υπάρχει ε, για να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα αυτό το θέμα και να το σπρώξουμε. Είναι ουσιαστικό θέμα, δεν θα πρέπει να γίνει κάτι που κάνουν κάποιοι με ρουτινιάρικο τρόπο, να χρησιμοποιήσουμε την ε, ορμή που υπάρχει αυτή τη χρονική στιγμή, το ζήλο που υπάρχει, το ενδιαφέρον και να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να το πάμε. Σε αυτή τη συνάντηση την 1η Μαρτίου να συγκρίνουμε επίσης ε, βέλτιστες πρακτικέ Ορισμένα έθνη, ορισμένα κράτη έχουν ε, πολύ χρήσιμε ιδέε για το εθνικό επίπεδο ή για μια περιφέρεια, ας πούμε, Φερρυπίν, οι σκανδιναβικές χώρες. συζητάνε πολλά για αυτά τα θέματα. Εκεί οι υπόλοιποι μπορούν να μάθουν από αυτές τις χώρες. Τρίτον, τρίτος άξονας, θα κοιτούμε το τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα. Τι μπορούμε να δώσουμε, να προσφέρουμε ε, για, στο, στη Σύνοδο το καλοκαίρι και στο ΝΑΤΟ. Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ε, αυτό είναι το δεύτερο, συγγνώμη, ε, ο δεύτερος άξονας ε, της ΠΕΣΚΟ και το, ο τρίτος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Πώς μπορούν να συνεργαστούν για τα θέματα αυτά οι δύο οργανισμοί. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, ότι μπορούμε να πετύχουμε εδώ μόνο να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμού. Στην ομάδα ad hoc υπάρχουν ε, ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και η Γενική Διεύθυνση MOVE και η Γενική Διεύθυνση TAXUD, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η UMS, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ελβετία. Όλοι ήταν παρόντε. Αυτή είναι μια συνταγή επιτυχία. Γιατί δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο μια χώρα, έναν οργανισμό. Ενδιαφέρει όλου. Έχουμε κοινά συμφέροντα εδώ και όλοι θέλουμε να σημειωθεί πρόοδο. Δεύτερον, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ένα θέμα που το ονομάζω χταπόδι μερικές φορές, γιατί έχει τόσα πολλά πλοκάμια, ε, δηλαδή πολλά θέματα εμπλέκονται εδώ, καταρχάς. Έχουμε τα εθνικά θέματα και έχουμε και τα διεθνή θέματα, έτσι πολύ σχηματικά και απλά. Το εθνικό σκέλος ε, πρέπει να έχουμε μια κυβερνητική προσέγγιση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να οργανώσουμε σε εθνικό επίπεδο όχι μόνο το Υπουργείο Άμυνα, μόνο, αλλά και το Εσωτερικών, ε, το Υπουργείο Υποδομών κτλ. Εν συνεχεία έχουμε θέματα τελωνιακά ή νομικά θέματα, τα οποία είναι ενωσιακή αρμοδιότητα και έχει σχεδόν 100% αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. εκει υπάρχουν εκει θέμα που είναι σε μια φαιά περιοχή, ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Κάποια θέματα είναι αμυγός εθνικά, κάποια αμυγός ενωσιακά και κάποια είναι υβριδικά. Η ιδέα λοιπόν είναι να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να πιέσουμε τις χώρες για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σε εθνικό επίπεδο και εν συνεχεία να πιέσουμε τα πράγματα ώστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χρειαστεί ατελείωτος χρόνος για να γίνουν απαραίτητες αλλαγέ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ελπίζουμε ότι ήδη φέτος το καλοκαίρι θα δείξουμε στους πολιτικούς μας ηθήνοντες ότι έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, όχι ότι έχουμε λύσει τα πάντα. Κάποια θέματα θα χρειαστούν χρόνια για να τα βελτιώσουμε και να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές, αλλά η φιλοδοξία μας είναι να έχουμε αυτά αποτελέσματα πρόθεσμα. Και μέχρι στιγμής είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα Αυτά και προσβλέπουμε στο μέλλον. Με εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ζαν Ιμαρτή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίε και κύριοι και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για την, την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της στρατιωτικής κινητικότητας ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και στην ατζέντα των κρατών μελών. Νομίζω ότι το σκηνικό έχει περιγραφεί αρκετά καλά, γι' αυτό και εγώ δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα στη σημασία που έχει αυτό το θέμα. Θα πω μόνο ότι δεν είναι νέο το θέμα αυτό. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, εργαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού άμυνας, για το σύστημα ανάπτυξης εδώ και πολλά χρόνια. Απλά την τελευταία χρονιά εμφανίστηκε πραγματικά πολύ ισχυρή πολιτική βούληση και η θέληση να επιταγηθούν οι εργασίες και να δοθεί ειδική προσοχή στο ζήτημα της στρατηγικής κινητικότητας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε και ο πρόσωπος του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζοντας βεβαίω και έχοντα κατά νου όλε τι εποχέ. όχι μόνο τι εποχέ πολέμου, τι περιόδου πολέμου και ενόπλων συγκρούσεων, αλλά και τι περιόδου ειρήνη. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια εξειδικευμένη ομάδα μελέτης από, την από, το, από τη Διευθύνουσα Επιτροπή του EDA για τη χαρτογράφηση των υπαρχουσών πρωτοβουλειών, την, ε, τον προσδιορισμό των ελλείψεων αλλά και με σκοπό να παρουσιαστούν στα κράτη-μέλη τα ευρήματα, τα πορίσματα όλης αυτής της διαδικασίας με συγκεκριμένους οδικού χάρτες που θα καθοδηγήσουν τα από εδώ και πέρα βήματα. Αυτή η ομάδα εργασίας δεν θα την χαρακτηρίζα ομάδα εργασία του, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα Είναι μια ομάδα εργασία που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, αλλά και εμπειρογνώμονες της ΕΙΕΔ, της Κομισιόν, Ταξούντ, ΜΟΥΒ την UMS και τη UMC. Πρόκειται δηλαδή για μια ομάδα εργασία στην οποία συμμετέχουν διάφορα μέλη τη ευρωπαϊκή οικογένεια και υπερβαίνει τα, τα στενά όρια μια απλή κοινότητα. Ε, Καθώ ε, ε, περιλαμβάνονται διάφορες, διάφορα θέματα. Ωστόσο, είναι πολύ συγκεκριμένη η εντολή που έχει λάβει αυτή η ομάδα εργασία από τα κράτη-μέλη. Συμμετέχουν και ε, ε, φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ προφανώς, έχουμε το MCCE, το European Transport Common, που θα συζητήσετε και αργότερα. Έχουμε και άλλους φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα εργασίας, προκειμένου να σκιαγραφεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και, μια, και να καταλήξουμε σε μια ορθή αξιολόγηση για το τι χρειάζεται να γίνει. Έπειτα από τέσσερις μήνες εντατικών εργασιών, η ομάδα εργασίας πλέον αναμένεται να ε, υποβάλει τους ε, οδικούς χάρτες σε τέσσερις τομείς με συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνουν και, συμπεριλαμβάνονται και οι, το ποιοι θα τεθούν επικεφαλής στον κάθε ε, τομέα. Τέσσερις λοιπόν είναι οι τέσσερις τομείς. που και το συνολικό έργο μας έχει έναν κοινό σκοπό. Βεβαίως να τονίσω ότι είναι λογικό όταν καθόμαστε μαζί και συζητούμε συγκεκριμένα θέματα να καταλήγουμε σε μια κοινή ανάλυση και σε κοινέ προτάσεις. Οι τέσσερις τομείς αυτοί είναι πρώτον η νομική διάσταση της ε, διασυνοριακής κινητικότητας Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ε, ενισχυθεί η συνέπεια μεταξύ των νομοθετικών επιπέδων, το εθνικό, το ενωσιακό και το διεθνές επίπεδο δηλαδή. όπου έχουν πλέον προσδιοριστεί και συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεύτερη διάσταση, δεύτερο τομέα μάλλον, είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με τα τελωνία. όπου έχουμε τον Ενωσιακό Τελεινικό Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2016 και είχαμε την ευκαιρία να εξορθολογήσουμε και να τυποποιήσουμε τις τελωνειακές διαδικασίες που ε, ακολουθούνται σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο προκειμένου να βελτιωθεί η ισχύουσα κατάσταση. Τρίτο τομέα είναι οι στρατιωτικέ απαιτήσει και υποδομέ. Πρόκειται ένα τομέα όπου το στρατιωτικό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η στρατιωτική επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούν στενότατα με το ΝΑΤΟ ε, είναι ένα θέμα το οποίο το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει αναδείξει ως εξαιρετικά σημαντικό και υπάρχει και σε αυτό το τομέα μια ισχυρή ε, διάσταση της διπλής χρήσης ε, όσον αφορά την, την, την σύνδεση, την, το συνδυασμό στρατιωτικών απαιτήσεων με μη στρατιωτικές υποδομές στην Ευρώπη. Και εδώ έχει σημαντικό ρόλο να παίξει η DG Move Τέταρτος τομέας αφορά τις ε, διασυνοριακές άδειες κινητικότητας. Αυτό είναι ο τίτλος αυτού του τομέα και είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε σε υπάρχουσες, σε ισχύουσες συμφωνίες. Υπάρχει ήδη ε, η τεχνική συμφωνία διαπίστευσης διπλωματών στην οποία συμμετέχουν 16 χώρες αλλά που προς το παρόν αφορά την αεροπορία. Σκοπός μας είναι να ενισχυθεί και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής με περαιτέρω συμφωνίες και να καλύπτει πλέον και τις οδικές ε, μεταφορές, τις θαλάσσιες, τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Σε σχέση με τα πορίσματα και τους οδικούς χάρτες που έχουν προταθεί, που θα παρουσιαστούν μάλλον στα κράτη-μέλη. Αυτοί, όπως σας είπα, θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο αφού η Διευθύνουσα Επιτροπή δώσει το πράσινο φως της και αυτή θα είναι η δική μας συμβολή ε, στη διαμόρφωση των ε, ενωσιακών σχεδίων δράσης ε, που αναμένεται να παρουσιαστούν το Μάρτιο. Η χαρτογράφηση των διαφόρων προβλημάτων που είναι το επίκεντρο της προσοχής αυτής της ομάδας εργασίας είναι απόλυτα απαραίτητη ακριβώς για να ενισχυθεί η συνειδητότητα, να ενισχυθεί ο συντονισμός, η συνέπεια, ε, μεταξύ των διαφόρων παικτών και φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και από αυτή την άποψη προφανώς πρόκειται μόνο για το πρώτο βήμα. Το επόμενο αποφασιστικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι να ε, δοθεί απάντηση στα πορίσματα στα οποία θα έχουμε καταλήξει και να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση. Από πλευράς λοιπόν του EDA, η Διευθύνουσα Επιτροπή θα προτείνει την εφαρμογή των οδικών χαρτών ε, με τις ε, ε, δραστηριότητες στις οποίες θα έχουμε καταλήξει. Μια άλλη συμβολή βεβαίως είναι το, το πρόγραμμα της ΠΕΣΚΟ, επικεφαλής του οποίου θα τεθούν οι κατοχώρες, γιατί η στρατιωτική κινητικότητα είναι μία από τις 20 δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ τα κράτη-μέλη. Άρα θα είναι σημαντική και η συμβολή μας σε αυτό το θέμα. Συμπερισματικά λοιπόν να πω ότι αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκα, περίπλοκο. Υπάρχουν διάφοροι φορείς, ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν από διαφορετικές αφετηρίες ο καθένας, γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρχει εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμός, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει και αν θέλετε προκειμένου να αγκαλιάσει ε, και φορείς και τομείς ε, της ζωής πλην της στρατιωτικής, να υπερβεί δηλαδή τα στενά όρια ε, των στρατών και με αυτά να δώσω το λόγο πίσω σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Πολύ σωστά τα όσα είπατε. Μας εξηγήσατε πάρα πολύ καλά τα διάφορα ζητήματα. Συνάδελφοι, μπορείτε να πάρετε τον λόγο. Κύριε ε, ε, Γκάλαρ, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε. Μας μάθατε πολλά. Το θέμα αυτό σίγουρα δεν είναι απλά σημαντικό χρήζει ήδη και πρακτικής εργασίας ήδη από τώρα. Δεν ξεκινάω από το μηδέν θα έλεγα. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι ευθυγραμμίστε παράλληλα με την ετήσια έκθεση της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας όπως το άρθρο 33 λέμε τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα συντονισμού της ταχείας μετακίνησης των αμυντικών δυνάμεων του προσωπικού, του εξοπλισμού και των προμηθειών για του σκοπούς τη κοινή πολιτική άμυνας, ε, ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο των ρητρών αλληλεγγύη, όπου όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αρρωγή και υποστήριξη ε, δύναμη του άρθρου 51 του Χαρτί των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, λέμε επίσης ότι απευθύνουμε έκκληση προς την Κομισιόν να προσιάσει ένα ουσιαστικό σχεδίο δράσης στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη μέχρι το Μάρτιο του 2018 το οποίο να συνάδει με τις σημερινές προσπάθειες εντός του ΝΑΤΟ. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν η Κομισιόν είναι σε θέση να τηρήσει αυτή την προθεσμία του Μαρτίου, αυτή την επιθυμία του Κοινοβουλίου για παρουσίαση ενός ε, πλήρους ενδελεχούς σχεδίου δράσης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Αναφερθήκαμε στην έκθεση αυτή πάλι. Λέμε ότι θεωρεί ότι η προτινόμενη Γενική Διεύθυνση Άμυνα θα πρέπει να έχει την ε, αρμοδιότητα να διασφαλίζει τα ανοιχτά σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση ε, προσωπικού και υλικού. Οπότε μήπως θα μπορούσε η Γενική Διεύθυνση μούβ ως κολαπτήριο αυτή τη στιγμή μέχρι να στηθεί η άλλη. Μήπως θα πρέπει να τη μετανομάσουμε γιατί η Γενική Διεύθυνση μου έχει και άλλες, ε, άλλα καθήκοντα. Δεν ξέρω πώς πάνε τα σχέδια για τη δημιουργία της DG Defense, γιατί αν παραμείνει στη MOVE, ορισμένοι μπορεί να προσβληθούν. Γιατί MOVE ε, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν ε, αφορά... Έχω και μια ερώτηση μάλλον που αφορά τη συγκεκριμένη δουλειά της μετακίνησης υλικού. Αυτό το θυμάμαι, αναφέρθηκε, θυμάμαι είχαμε μια πλήρη κάλυψη στη δύση όλων των γεφυρών και των μικρών. Τις γνωρίζαμε όλες, θυμάμαι, αυτές τις πινακίδες ε, στρατιωτικού φορτίου σε κάθε, ακόμη και στη μικρότερη γέφυρα, ώστε ο κάθε οδηγός ε, φορτηγού ε, άρματος να γνωρίζει αν μπορεί να διέλθει ή όχι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα. Ε, δεν θα έπρεπε λοιπόν να συντάξει κάποια νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπό τη μορφή ενό κανονισμού. Γιατί χρειαζόμαστε ομοιομορφία σε αυτά τα θέματα. Χρειαζόμαστε ομοιόμορφε πινακίδε και σήμανση που να μα λέει ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι μια συγκεκριμένη προθεσμία και να μα λέει ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε κάποια στιγμή τέτοια εναρμονισμένη, ομοιόμορφη ε, επισήμανση μέσω αυτών των πινακίδων, των στρατιωτικών πινακίδων. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ε, θα βοηθούσε ιδιαίτερα τη μετακίνηση των στρατευμάτων. Και η άλλη πτυχή που αναφέρθηκε, όσον αφορά αυτή τη διασυνοριακή μετακίνηση των στρατευμάτων, ε, εν συντομία το λέμε στρατητικό Σέγγεν, στρατιωτικό χώρο Σέγγεν. Ε, και αυτό χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Το θυμάμαι, διότι είμαι και κάποιες ηλικίε ότι παλιότερα όταν είχαμε λιγμούς του ΝΑΤΟ έρχονταν οι Αμερικάνοι δεκάδες χιλιάδες περνούσαν τον Ατλαντικό και δεν νομίζω ότι όλοι καθόντουσαν να αναδείξουν τα διαβατήριά του ε, για να σφραγιστούν τα διαβατήριά του στα σύνορα. Η διαδικασία ήταν αρκετά γρήγορη αυτή τη διέλευση των σύνορων το παλιό καλοκαιρό. Και τώρα στην Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις νομοθετικές αρμοδιότητες που έχουμε, πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αυτό το στρατιωτικό χώρο Σέγγεν για το προσωπικό, για το στρατιωτικό προσωπικό, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε. Και το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω είναι ε, αν λάβουμε αυτή την ε, ενδελεχή έκθεση από την Κομισιόν ε, μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ή κάποια στιγμή αργότερα δεν θα πρέπει να γράψουμε στα πρακτικά μας έντε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτήν την έκθεση διότι εγώ γνωρίζω και ότι υπάρχει και μια άλλη επιτροπή που λόγω ε, του ότι δεν έχει πολλή δουλειά σκέφτεται να μας την αρπάξει ενώ θα πρέπει εμείς να είμαστε η καθουσία αναρμόδια αρμόδια επιτροπή ε, μόλις έρθει η έκθεση από την Κομισιόν Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε Ευχαριστώ ιδιαιτέρως ε, τους παρόντες. Μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο. Ε, μια ανακοίνωση που προέβλεπε τη δυνατότητα ε, εκ μέρους της ΑΦΕΤ μάλιστα έχει ζητηθεί να απαντήσουμε σε αυτό το έγγραφο. Με ένα έγγραφο το οποίο να μας προετοιμάζει αυτό το σχέδιο δράσης. Σχέδιο δράσης που αναμένουμε, διότι σίγουρα καλό είναι να έχουμε λάβει ε, τα κείμενα καιρό πριν, όταν αυτά τα κείμενα προκαλούν μεγάλες συζητήσεις. Έχω μια ε, ερώτηση προς τον Δόκτωρ Μόλενάρ. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που κατά κάποιο τρόπο πάντα ε, συναντά μπροστά μας το Brexit. Ε, έχουμε συζητήσει τι θα γίνει, πώς θα επηρεάσει το Brexit τα σχέδιά μας. Διότι όταν μιλάμε για υποδομές, ε, δεν μιλάω για υποδομές κοινέ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ίσως ήδη να συζητείτε κάπου. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για το έγγραφο που έδωσε. Αλλά πιστεύω ότι τα σημαντικά πράγματα είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να στραφούμε προς τη Γενική Διεύθυνση MOVE και άλλους διευθυντές και να προσπαθήσουμε να τους δείξουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε την κινητικότητα φυσικά τώρα διότι μιλάμε και μετακίνηση προσωπικού Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα προετοιμάσουμε. Όλη αυτή την κινητικότητα πρέπει να την προετοιμάζουμε σε εποχές ειρήνης. Διότι προφανώς πρέπει να συντηρούμε τις υποδομές, να τις βελτιώνουμε, να τις ενισχύουμε σε κάποιους τομείς. Και μετά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση... Τι ιδέα έχετε για το πώς θα σχεδιάσουμε αυτό το, αυτή τη χρηματοδότηση. Ε, έχουμε κάνει λόγο πολύ για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τις κατεπίγουσες ανάγκες που έχουμε για χρηματοδότηση που συνδέονται με τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την προσθεμένη αξία που μπορεί να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να τις προωθήσουμε. Λοιπόν, για τις ε, υποδομές λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ε, σε σχέση με την ασφάλεια, από τη μία, αλλά από την άλλη και το επιχειρησιακό κομμάτι. Ε, χρειαζόμαστε πλοία, χρειαζόμαστε τρένα, χρειαζόμαστε αεροπλάνα για να μετακινήσουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τον κλάδο για να δούμε πώς θα τους μετακινούμε αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Κώστερ, εσείς δεν, δεν έχετε σχεδιασμό, δεν έχετε χάρτες ε, Πώς σχεδιάζετε την ε, συνεργασία. Θυμάστε την επιχείρηση Αταλάντα. Κάποιος είχε πει ότι η Αταλάντα είναι το προανάκρουσμα μιας στρατιωτικής επιχει... Ε, επιχειρησιακής ικανότητας. Ε, τι, ποια είναι τα θετικά στοιχεία Τη Αταλάντα που θα κρατήσετε για να αναπτύξετε κάτι τέτοιο σε μεταγενέστερη φάση. Επίση, μας, μιλήσε, κάποιο ομιλητή για μια συζήτηση που κάνουν τα σκανδιναβικά κράτη. Πώ μπορούμε να ε, μεταφέρουμε το μοντέλο αυτό ε, στο Νότο και στην Ανατολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι. Γιατί εμεί ε, στο Νότο είμαστε στην ε, πρώτη γραμμή του πυρό. και είναι σημαντική η συνεργασία. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αγιαλά Σέντερ. Ήθελα και εγώ ως τακτικό μέλος της Επιτροπής να κάνω μια ερώτηση. Μια παρατηρήσή μου είναι ότι κατά καιρούς, ακόμη και σήμερα, χρησιμοποιούμε τον όρο ε, στρατιωτικός χώρος έγκεν». στρατιωτικό Σέγγεν. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον ΝΑΤΟ ακούσαμε σχόλια από ε, τον κύριο Ιαν Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και μας ζήτησε να μην χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Και νομίζω ότι είχε δίκιο. Διότι Υπάρχουν και ευκολότεροι τρόποι βελτίωσης της κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα στρατεύματα που μας ε, υπερασπίζουν, όχι μόνο που μας προστατεύουν, όχι μόνο για λόγους κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, αλλά και για καθαρά αμυντικούς λόγους. Και όλο αυτό εντός ε, του πεδίου αρμοδιοτήτων του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρθηκε σήμερα πριν από μερικές ώρες ε, από τον ε, πρόεδρο της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος μας είπε ότι ενώ οι κυρίες δραστηριότητες τους είναι περισσότερο προστασία όταν μιλάμε για να αποφεύγουμε τη διπλή δουλειά η άμυνα αποτελεί σε μεγαλύτερο βαθμό αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ Καθημερινά όμως ακούμε διάφορες ε, δηλώσεις ε, και μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Γιούγκερ για την ε, Αμυντική Ένωση. Η ερώτησή μου λοιπόν την απευθύνω κύριε στον Διευθυντή Κώστερ και στον Διευθυντή Ρέιτερς και πιθανώς και προς τον κύριο Μαρτί. Θα πρέπει να βρούμε μια άκρη για αυτό το ζήτημα και να δούμε και ποιες είναι οι προοπτικές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε νέες οδούς ε, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να φέρουμε στρατεύματα εξωτερικά, δηλαδή από κράτη που δεν είναι, από κράτη μέλη, δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ενδεχομένως από το Ηνωμένο Βασίλειο, από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, αμερικανικές, καναδικές, που ήδη ε, έχουν ε, αναπτυχθεί στην Ευρώπη, βρίσκονται στην Ευρώπη, στα κράτη της Βαλτικής, ε, στη Ρωμανία, στην Πολωνία και αλλού. Και φυσικά λαμβάνω και υπόψη και τη διάσταση της παρουσίας του ΝΑΤΟ εκεί. Και τη... λαμβάνω υπόψη και την ανάγκη να ενισχυθεί η κινητικότητα. Ποιες είναι οι απόψεις γι' αυτό. και ειδικότερα όσον αφορά αυτά τα ζητήματα της διπλής χρήσης. όπου ορισμένα ζητήματα είναι καθαρά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άλλα καθαρά των κρατών μελών. Αγαπητοί κύριοι, λοιπόν, έτσι όπως κάνετε τις παρουσιάσεις σας, ε, ε, ξαναπάρτε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γκάλλερ θέλει ξανά το λόγο. Ναι, εν συντομία, Νομίζω ότι εσκεμένα καλέσαμε και τους δύο οργανισμούς. Γιατί, διότι εδώ τίθεται θέμα συμπληρωματικότητας. Δεν θέλουμε δηλαδή να, να μάθουμε την αρμοδιότητα, την αποκλειστική του ενό ή του αλλονού, αλλά τη συμπληρωματικότητα. Δεν έχει νομοθετική εξουσία το ΝΑΤΟ, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε εσωτερικά τα σύνορα και καθοριζώντας τους λόγους. Το έχουμε κάνει για αγαθά, για πρόσωπα και στο μέλλον μπορούμε να το κάνουμε για στρατεύματα, για να διευκολύνουμε ουσιαστικά την κατάσταση. Δεν μιλάμε τώρα μόνο προ εμά νομοθετικά, μιλάμε και στον κόσμο και στου λαού μα. Ξέρουν τι σημαίνει το Σέγγεν, ξέρουν τι θέλουμε να επιτύχουμε πολιτικά. Οπότε και τα στρατεύματά μα για οποιοδήποτε σκοπό, για ελιγμού ή για οποιαδήποτε ζητήματα πραγματικά αμυντικά θα πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα. Γι' αυτό το λόγο αναφέρω εσκεμένα αυτό το θέμα, παρότι δεν φαίνεται να υπάρχει νομικό κείμενο, αλλά για να το κατανοήσουμε όλοι. Ο κόσμο, ε, γι' αυτό το ονομάζω εγώ έτσι, γιατί ο κόσμο καταλαβαίνει τι θα πει Σέγγεν, γι' αυτό αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορούμε να το μεταφέρουμε και στη στρατιωτική σφαίρα. We start with uh, answers of Director Molinar. Να ακούσουμε τώρα τι απαντήσει του Διευθυντή του κ. Μολινάρ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλε αυτέ τι ερωτήσει. Για το στρατιωτικό Σέγγεν, Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς έτσι με λίγα λόγια. Το κρίσιμο όμως που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε, ε, χρειαζόμαστε ταχεία κινητικότητα και μεταφορά, όχι απλώς ελεύθερη. Να επιταγηθούν δηλαδή διαδικασίες ελέγχου κατά την ε, διέλευση των συνόρων όχι να μην υπάρχουν καθόλου έλεγχοι, απλά να ε, μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε και να απλοποιήσουμε τι διαδικασίες προκειμένου να, επιταχυνθεί, να επιταχυνθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι το, το βασικό σημείο που, κρατήσει να, που αξίζει να κρατήσουμε. Γι' αυτό και στο παρελθόν είχαμε πει να εγκαταλείψουμε αυτή την έννοια του στρατιωτικού Σέγγεν που μπερδεύει, συσκοτίζει τα πράγματα για το σχέδιο δράσης που καταρτίζει η Κομισιόν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με ειδική ε, ε, ευθύνη της DG Move. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση και τώρα και έχουμε συλλέξει και τις απόψεις των, ε, των κρατών μελών, των εμπειρογνωμόνων αυτό που απομένει να γίνει είναι να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράση, όπως είπα θα γίνει το Μάρτιο. Για την Γενική Διεύθυνση Άμυνα δεν θα επισέλθω εγώ, θα τα αφήσω σε όλους Για το Brexit ήταν ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Για να μην ειλικρινείς, οι συζητήσεις για τον Brexit βεβαίω κατ' εξισοχήν ε, διεξάγονται σε άλλο πλαίσιο. Γενικά όμως μπορώ να πω και αυτό είναι το βασικό αίσθημα που επικρατεί στη συζήτηση, είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε <clears throat> ότι θα σημειωθεί πρακτική πρόοδος και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Το τόνισε και η πρόεδρος αυτό. Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και βεβαίως ακολουθώντας τις ε, καλύτερες δυνατές διαδικασίες για να προχωρήσουμε. Ένα Γρήγορο σχόλιο για το Αταλάντα που είναι ναυτική επιχείρηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σομαλία βέβαια, από αυτή την άποψη δεν σχετίζεται ακριβώς με το σημερινό θέμα συζήτησης που είναι στρατιωτική κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, στόχος αυτής της ναυτικής επιχείρησης είναι μεταξύ άλλων και η προώθηση της, ε, της ε, κινητικότητας, της ελεύθερης μεταφοράς ε, εμπορευμάτων και ανθρώπων. Ε, άρα από αυτή την άποψη δεν άπτεται ακριβώς αυτό του θέματος της στρατιωτικής κινητικότητας εντός Ευρώπης, ε, της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά σημειώνω αυτά που είπατε και πρέπει να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την καλύτερη δυνατή προστασία των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διεθνώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τη συνεργασία του Δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, ε, συμφωνώ και εγώ ότι ο ρόλο των δύο οργανισμών είναι συμπληρωματικό ε, από πολλέ απόψει σε πολλού τομεί. Στην πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μέσα και εργαλεία τα οποία μπορούμε βεβαίω και εμεί να συνεισφέρουμε και σε τελική ανάλυση αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα αυτά βοηθούν τα κράτη-μέλη. 22 από αυτά ε, μάλιστα συμμετέχουν και στους δύο οργανισμούς, άρα ε, βεβαίως προς όφελός τους είναι να εξασφαλιστεί καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, βάσει πάντοτε των ε, σωστών αξιών και αρχών, όπως πάντα. Κύριε Ρόιτερς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι αυτό το σχέδιο δράσης τώρα να είναι έτοιμο το Μάρτιο. Ε, υπάρχει κοινή ανακοίνωση. Είναι πολύ σημαντικό λόγω των σημαντικών εξελίξεων που θα έχουμε το, την Άνοιξη και το καλοκαίρι. Τώρα, ποια γενική διεύθυνση θα είναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Το βασικό είναι να συνεργαστούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να δώσουμε αποτελέσματα με το σχέδιο δράσης και μετά μέσα στο 2018. Κύριε Γκάλερ, μιλήσατε για τα στρατιωτικά θέματα, τα οποία εντοπίζουμε μαζί με την UMC, ε, με την EDA και το ΝΑΤΟ. Ε, και θα πρέπει το στρατιωτικό σκέλος να συμβατώ με το μη στρατιωτικό σκέλος, το πολιτικό σκέλος δηλαδή, ούτω ώστε να, πάρουμε, να λάβουμε υπόψη μας και τον κονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, Από την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για, τον, το στρατιωτικό σκέλος ε, που θα ήταν χρήσιμο και για το πολιτικό σκέλος και θα τα βάλουμε στον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Είναι σημαντικό να βελτιστοποιήσουμε την διτή χρήση, το dual use. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Αγιάλα Σέντερ, αυτή η ανάλυση, όπως ξέρετε, είναι εν εξελίξη. Έχουμε καταρχάς το εργαλείο διευκόλυνση για την διασύνδεση της Ευρώπης ε, και τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και είναι σημαντικό πώς θα χρηματοδοτήσουμε. Καλό είναι ε, να έχουμε και την στρατιωτική γνώση παράλληλα. Ε, αν βάλουμε 24 εκατομμύρια στο TNT, καλό είναι να το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο με βάση και την γνώση στο στρατιωτικό σκέλος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας ε, ε, εμείς, ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή τη χρήση. Τώρα, για το αν οι επενδύσεις αυτές χρειάζονται κάποια κονδύλια, θα το δούμε. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το Connecting Europe Facility μας λέει ότι το μοντέλο αυτό ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και θα μπορούσε να είναι, χρήσιμο, να είναι χρήσιμο και αργότερα όταν ε, εντοπίσουμε τα προβλήματα και μετά περάσουμε στην εφαρμογή. Να μην τα κάνουμε ανάποδα. Φυσικά ο κύριος Κώστερ θα μιλήσει για το τροχαίο υλικό. Ε, εγώ μίλησα περισσότερο για τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη και για το TNT. Ε, ευχαριστώ, Διευθυντή ο κ. Κώστερ. Υπάρχουν δύο θέματα, δύο ερωτήσει που μου υποβλήθηκαν ευθέω. Καταρχά, η άσκηση χαρτογράφηση. Δεν κατάλαβα τη σχέση με την επιχείρηση Αταλάντα. αλλά και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αμερικανών έχουν υποδομές, ε, βάσεις δεδομένων, ατελείς όμως. Γι' αυτό λοιπόν, καθώς και η, Αμερικανική, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση καθώς και η Αμερικανική Διοίκηση. Πρέπει να, δούμε τι ξέρει ο, άλλ, ο άλλος, ο εταίρος μας, ας πούμε, αντί να ξεκινάμε από το μηδέν. Ένα από τα πρώτα βήματα λοιπόν για να καταλάβουμε ε, ποια είναι η κατάσταση των υποδομών είναι να πάμε να συνομιλήσουμε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι επίσης έχουν βάση δεδομένων και να δούμε αν μπορούμε να συμπληρώσουμε τις γνώσεις που έχουμε. Ε, αν μπορούμε να προχωρήσουμε δηλαδή εκεί. Τώρα, για το στρατιωτικό Σέγγεν, ακούσατε γιατί ο όρος αυτός ε, προκαλεί σύγχυση, να προσθέσω ότι για πολιτικούς λόγους καλό θα ήταν πιο επικοδομητικό να βρούμε ένα νέο πιο ουδέτερο όρο παρά να ζητούμε από μια οργάνωση να <laughs> υιοθετήσει τον όρο που χρησιμοποιεί ένας, μια άλλη οργάνωση. Έτσι. Είναι πολιτική, πολιτικός ρεαλισμός αυτό. Η... Σε ό,τι αφορά τους καονισμους να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος. Εμείς στο ΝΑΤΟ δεν έχουμε ακριβώς νομοθεσία, αλλά έχουμε διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες. Φερρυπίν, η επιχείρηση ISAF, η οποία ε, αναπτύσσεται εδώ και 10 χρόνια. Χρησιμοποιεί μια μορφή αδειοδότησης αγαθών, το F302, έτσι λέγεται αυτό το έντυπο, δεν το χρησιμοποιούν μόνο οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, αλλά όλοι οι εταίροι, 25 χώρες και πλέον που συμμετέχουν στην ISAF. Όταν μιλάμε για μία, ε, ένα έντυπο ή μία άδεια, ας πούμε, για να μεταφέρουμε, να πάρει άδεια, ας πούμε, η μετακίνηση στρατιωτικού υλικού στην Ευρώπη, ε, καλό είναι να δούμε τι υπάρχει παρά να ξεκινάμε, ας πούμε, από το μηδέν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι δεν μιλάμε για νομοθεσία απλώς για τη διαλέψη των σύνορων. Ε, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Υπάρχουν και άλλα πολύ περισσότερα θέματα, κανόνες κτλ. Ε, και υπάρχουν και άλλα προσκόμματα που δεν βοηθούν ε, την ε, μετακίνηση στρατιωτικού υλικού. Παραδείγματο χάρη ε, στη Γερμανία τα φορτηγά δεν μπορούν να μετακινούνται το Σαββατοκύριακο. Το Επίσης, ε, επιτρέπεται ένα ρημουλκό ενός φορτηγού να μετακινείται εντός της εβδομάδας μόνο το βράδυ, ανάμεσα στις 12 και στις 6 το πρωί, 12 το βράδυ και στις 6 το πρωί. Ε, μια δεξαμενή, ας πούμε, σε ένα φορτηγό. Και αυτά εν καιρό ειρήνης. Έτσι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την νομοθεσία μόνο και μόνο γιατί έχουμε μια άσκηση, να γυμνά, κάποια γυμνάσια, πούμε. Αλλά μια, μια χώρα όπως η Γερμανία που είναι στη μέση της Ευρωπαϊκής Υπήρου θα πρέπει να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Ε, και να σας πω και κάποιο, κάτι που τα περιπλέκει τα πράγματα. Μερικές από αυτές τι αρμοδιότητες δεν είναι καν ομοσπονδιακές. Είναι ε, αρμοδιότητες των Λέντερ. Ζητώ συγγνώμη που τώρα ονοματίζω τη Γερμανία. Ε, δεν μιλάμε για νομοθεσία απλώς μας επιτρέπει να περάσουμε στην διέλευση των συνόρων, να λύσουμε αυτό το θέμα, να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, ο Διευθυντής κ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, επί του τελευταίου αυτού σημείου και για να δώσω και κάποια παραδείγματα από την Ολλανδία, για μας ε, δεν είναι μόνο η κεντρική αρμοδιότητα των ε, Υπουργείων αλλά και η αρμοδιότητα του Δημαρχού του Ρότερνταμ για παράδειγμα ο οποίος έχει δικές του αρμοδιότητες η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι έχει δικές της ε, αρμοδιότητες οπότε δεν μιλάμε μόνο για την κεντρική κυβέρνηση αλλά και για τις τοπικές Όσο πιο πολύ λοιπόν το ψάχνει κανείς τόσο πιο πολύπλοκο διαπιστώνει ότι είναι όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλες τις χώρες μας. Έγινε μία ερώτηση για τις βόρειες χώρες. Νομίζω ότι ορισμένα κράτη... Ξέρετε, έχουμε κάνει συζητήσει σε ομάδε εργασία και βλέπει κανεί παραδείγματα ορισμένων χωρών. Σε ορισμένε χώρε τα πράγματα οργανώνονται καλύτερα από τι άλλε. Αυτό είναι απλά γεγονό. Σε ορισμένε χώρε ε, υπάρχει περιφερειακή συνεργασία, όπω η συνεργασία των ε, βόρειων χωρών, όπου συζητούν ήδη τα ζητήματα αυτά και εκεί μπορεί κανείς να αποκομίσει πολύ ενδιαφέροντα διδάγματα. Και αυτό θα κάνουμε, ελπίζουμε, στη συνάντηση της ΠΕΣΚΟ, να αξιοποιήσουμε τα έξυπνα παραδείγματα, τις βέλτιστες πρακτικές και να δούμε πώς ε, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και σε άλλες χώρες. Επίσης, ε, τίθεται και το άλλο ερώτημα, υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει από όλες τις πλευρές πολιτική βούληση Οπότε όταν μιλάμε για αυτή την έκθεση υπάρχει ευελιξία από όλες πλευρές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις της ΠΕΣΚΟ για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βούληση αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη τη ΠΕΣΚΟ, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. ειδική σα επιτροπή. Μπορείτε να κάνετε προσπάθειε για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη πολιτική βούληση για να επιληθούν τα διάφορα ζητήματα τα οποία διακυβεύονται. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Μαρτί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για όλε τι ερωτήσει. Φυσικά δεν θα μπω στη συζήτηση με όλα αυτά τα ονόματα. Το θέμα είναι ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας που θέλουμε να ορίσουμε για όλο αυτό. Προφανώς εδώ στη συζήτηση η αίσθηση που αποκτώ από τα κράτη-μέλη είναι ότι ο στόχος εδώ φυσικά δεν είναι να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τις στρατιωτικές τους ε, δυνάμεις που, τις δυνάμεις που θα μπαίνουν στην επικράτειά τους. Δεν θέλουμε να τους αφαιρέσουμε δηλαδή δυνατότητα ελέγχου, αλλά απλά όταν λαμβάνεται μια απόφαση σε πολιτικό επίπεδο να μπορούν τα πράγματα να κινηθούν γρήγορα, να μην υπάρχει κάτι που να τις εμποδίζει, ε, κάτι που να εμποδίζει την απλή υλοποίηση της πολιτικής απόφασης η οποία θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα, γρήγορα, ομαλά. Αυτά όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας. Όσον αφορά την υποδομή, τις υποδομές, αυτό νομίζω είναι στόχος του τρίτου τομέα που περιγράψαμε. Το να υπάρχουν σαφείς απαιτήσει. Αυτό υπόθηκε ήδη. Σαφείς απαιτήσει του στρατιωτικού σκέλους ώστε οι πολλοί και διάφοροι επενδυτές ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις λαμβάνοντας αυτές τις απαιτήσει υπόψη όχι να γίνονται αυτέ οι επενδύσεις μετά από την κρίση λόγω έλλειψης γνώσεων ε, ξαφνικά να καταλήγουμε σε κάτι ελλειπέ. Αυτό μας οδηγεί απευθείας ε, και στο ζήτημα των επενδύσεων. Πιστεύω ότι εδώ, επειδή το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, υπάρχει προφανώς ανάγκη να καθοριστούν όχι μόνο οι απαιτήσει αλλά και οι επενδύσει και να βρεθεί ο κατάλληλο τρόπο συνδυασμού των διαφόρων τύπων επενδύσεων από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ. με τη χρήση των κατάλληλων ε, νόμων, ε, νομοθετικών μέσων για όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα του συνδυασμού των επενδύσεων από διάφορε πηγέ ε, που εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε έναν εξελισσόμενο κόσμο. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα για την Αταλάντα που ίσως δεν σχετίζεται άμεσα με το επίκεντρο του ζητήματος της κινητικότητας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που σε κάποιο βαθμό σχετίζεται όμως όταν λέτε τέτοια σχόλια θυμήθηκα θυμήθηκα ότι μία από τις προτελεότητες ανάπτυξης ε, δυνατοτήτων που συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη ήταν να συμφωνήσουμε θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά μία ε, δυνατότητα θαλασσιπητήρησης ε, για τις νάρκες, για το, το επίκεντρο λοιπόν του ζητήματος που θέλουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε με τη στρατηγική κινητικότητα είναι ότι υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες ε, των κρατών μελών που μπορεί να γίνουν με συμμετοχή ε, των επιμέρους χωρών όπως ε, η, αερομετα... η αεροδιακομιδή, για παράδειγμα, οι αερομεταφορές ε, και με τις σχετικές επενδύσεις. Τώρα όσον αφορά τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν ε, το πνεύμα της εργασίας μας ε, είναι να έχουμε και εξωτερικούς συμμετέχοντες. Αυτό συζητάμε. Το να έχουμε τις ΙΠΑ στις συζητήσεις μας για την Ελβετία, εταίρους μας ε, που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τελικά το αποτέλεσμα να είναι επωφελές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για όλους τους συμμετέχοντες. Προφανώς και αυτός είναι ο σκοπός μας, ε, να μην έχουμε αποκλεισμούς, ε, να βελτιστοποιούμε τα ωφέλη. Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θα πρότεινα να ολοκληρώσουμε 12.30 ώρα ακριβώς την συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε για να ανταλλάξουμε απόψεις στο θέμα της στρατιωτικής κινητικότητας. Θα δοθεί συνέχεια, συνέχεια βέβαια. Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και θα εξετάσουμε από κοινού ή το καθένα ξεχωριστά διάφορα θέματα που θα ανακύπτουν κατά την πορεία της κατάρτισης του οδικού χάρτη προκειμένου να φωτίσουμε τα θέματα αυτά από όλες τις ε, πλευρές. Ένα χειροκρότημα για τους ομιλητές μας, παρακαλώ. Uh, 2.30. Ξαναρχίζουμε στις 2.30. Done. Διαδικαστικό θέμα. Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσατε να προτείνετε να κάνει κάτι και η, υπο... να κάνει κάτι και η υποεπιτροπή μας να ετοιμάσει ένα ψήφισμα ή μια προφορική ερώτηση ή έστω μια γνωμοδότηση για την ανακοίνωση αυτή για να συνεισφέρουμε και εμείς το σχέδιο δράσης για να ξεχερσώσουμε πούμε, το έδαφος για να ετοιμάσουμε το σχέδιο δράσης. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε, αλλά νομίζω θα ήταν χρήσιμο. για να προετοιμάσουμε και τους συναδέλφους για τη συζήτηση αυτή. Δεν ξέρω αν γίνεται. Βεβαίω. ακούμε τη συμβουλή σας, θα τη λάβουμε υπόψη, ε, θα το δούμε η γραμματεία και οι συντονιστές για να δούμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε και να το προτείνουμε. Παρακαλώ. Δυόμιση η ώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που επίσης είναι πολύ σημαντικό.